Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο κύριο Κατάινεν στην ε, Επιτροπή μας, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συζητήσουμε το πρόγραμμα δράσης για την κυκλική οικονομία ε, στις 16 Μαρτίου Μαρτίου του 2016 είχαμε ζητήσει μια ενημέρωση και θα θέλαμε τώρα να ε, ενημερωθούμε για τις εξελίξεις σε σχέση με την ε, προηγούμενη επίσκεψή σας, όπως επίσης ε, θέλουμε να δούμε τι γίνεται και με την δημοσίευση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο, με, την, με τη δράση για την κυκλική οικονομία. Ήδη ε, είχαμε αποφασίσει να ζητήσουμε από τον Αντιπρόεδρο ή από εσά να έρθετε εδώ να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και σας ε, δίνουμε τον λόγο καταρχάς και μετά θα υπάρξει και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Το σημερινό θέματα, θέμα μας είναι η κυκλική οικονομία που είναι πολύ επίκαιρο θέμα διότι έχουμε δημοσιεύσει σήμερα ένα κατάλογο προϊόντων μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για το eco-design. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα αργότερα στην ομιλία μου. Αλλά πραγματικά ε, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε στην ε, κυκλική οικονομία. Πολλοί από εμά ε, συμφωνούν ότι η κυκλική οικονομία αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μετάβαση από την γραμμική οικονομία στην κυκλική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι τα σχήματα κυκλικής οικονομίας υπάρχουν ήδη στην αγορά, απλώς είναι πιο παραγωγικά και, προς, ε, και προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ότι η γραμμική οικονομία, από στη γραμμική οικονομία. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται και η χρηματοδότηση, μπορούμε με τον τρόπο αυτό να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα και την κοινωνική μας πολιτική. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επομένω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η κυκλική οικονομία. Είμαστε στο σωστό δρόμο, πιστεύω, και πηγαίνουμε καλά, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση του πακέτου κυκλικής οικονομίας. Πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν έχει αρχίσει να εφαρμόζει ε, το σχέδιο δράσης με έναν σταθερό ρυθμό και έχουμε υποβάλει και τις νομοθετικές προτάσεις για τις online πωλήσει προϊόντων και, ε, και τις ε, προτάσεις για, τα, για τις εγγύησεις των προϊόντων επίσης. Πάλι και αυτές οι νομοθετικές προτάσεις. Επίσης, Υπάρχει και η πρόταση για, την, ε, για, τον, αναθεωρημένο κανονισμό για τα ε, λιπάσματα, όπως επίσης και για τις ε, ε αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές. Η Κομισιό θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη της εφαρμογής ε, του σχεδίου δράσης μέχρι το Γενάρη του 2017 και ε, θα υπάρξει και μία ανακοίνωση για τα, που αφορά τα, τα απόβλητα στην ενέργεια. Ταυτόχρονα ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε και μία πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας. Τώρα, οδηγία eco-design. το eco-design είναι ένα ε, ζωτική σημασίας ε, ε, εργαλείο για να αποκτήσουμε την κυκλική οικονομία, γιατί δημιουργεί και κίνητρα, αλλά και ένα πεδίο ισότητας για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα και που εισάγουν προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι παραπάνω από ένα project εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα, ένα πεδίο και για την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών προϊόντων αλλά και των εισαγωμένων προϊόντων. Πρέπει να το δούμε το eco-design από τρεις πλευρές. Από, την, από πλευρά των καταναλωτών, τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές δηλαδή. Δεύτερον, να δούμε τι, τα πράγματα από την οπτική γωνία της βιομηχανίας και τρίτον το από τα αποτελέσματα σαν αποτέλεσμα του eco-design να μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ας κάνουμε μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά τους καταναλωτές. Μειώνουμε την την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στα χέρια των κυβερνήσεων ή των ε, ε, όσων αποφασίζουν για τις πολιτικές. Αυτό εξαρτάται και από τους καταναλωτές όταν καθημερινά επιλέγουν κάποια προϊόντα. Και όσο πιο εξουσία, αν θέλετε, ή δύναμη έχουν οι πολίτες, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες να εξυγχρονιστούν. Η οδηγία για το eco design είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους καταναλωτές και με τον τρόπο αυτό να μπορούν οι πολίτες να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής, οι οργανώσεις Ευρωπαίων καταναλωτών μάλλον, θα έλεγα, ότι ε, υπολογίζουν ε, τις ε, οικονομίες των νοικοκυριών στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι 450 ευρώ το χρόνο. Η Κομισιό θεωρεί ότι η οικονομία που μπορεί να πετύχει ένα κλασικό νοικοκυριό στην Ευρώπη φτάνει τα 500 ευρώ το χρόνο. Επομένως, οι συνειδητοποιημένες επιλογές ε, μπορούν να εξοικονομήσουν ένα σημαντικό ποσό για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Τώρα, ας δούμε την κατάσταση από πλευρά των επιχειρήσεων. Το eco-designing και η σήμανση eco-design μπορεί να βοηθήσει, διότι ορίζει ομοιόμορφα πρότυπα, προστατεύει το περιβάλλον και επίσης προωθεί τις α, επενδύσεις σε νέα προϊόντα και σε καινοτόμες λύσεις. Το πλαίσιο του eco-design, σύμφωνα με τις μελέτες, ε, λέει, λέει, προβλέπει τέλος πάντων ότι μπορεί να εξοικονομήσει 55 δισεκατομμύρια για την ε, βιομηχανία ετησίως. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι βιομηχανίες καταναλώνουν ενέργεια. Η κατάσταση επομένω είναι win-win και από πλευρά τη βιομηχανία και από πλευρά των καταναλωτών. Αυτό όμως δεν αφορά και για τα, τα ιδεατά προϊόντα, αν θέλετε, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια, για εκατομμύρια προϊόντων, προϊόντων που επηρεάζουν ένα νοικοκυριό. Αυτή τη στιγμή Ε, από την αρχή της ε, οδηγίας για το eco-design έχουμε υπολογίσει ότι εξοικονομούμε ενέργεια που ε, αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενέργειας της Ιταλίας για έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα, βέβαια πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω δουλειά, περισσότερο Ε, αποδοτική έτσι ώστε το 2030 να έχουμε εξοικονομήσει που παραπάνω ε, από αυτή που έχουμε τώρα που να αντιστοιχεί με την ετήσια κατανάλωση της Σουηδίας. Δηλαδή να έχουμε την ε, κατανάλωση της Ιταλίας και της Σουηδίας μαζί ως οικονομία. Όπως σας είπα, σήμερα δημοσιεύσαμε ένα κατάλογο προϊόντων που θα προσθεθούν ε, στα προϊόντα του Eco Design. Έξι, προ, έξι κατηγορίες πολλές ε, ανελκυστήρες, ε, ηλιακά πάνελ και τα και όλα αυτά τα εξαρτήματα αν θέλετε και έχουν επιλεγεί λόγω του, των δυνατοτήτων που προσφέρουν δεν είχαμε καμία, κανένα, καμία πολιτική διαπραγμάτευση, τέλος πάντων, ε, η παζάρι, ε, με επιστημονικά κριτήρια έγινε η επιλογή. Δηλαδή, εάν η πρόταση αυτή προχωρήσει, με λίγα λόγια, οι Ευρωπαίοι θα έχουν ε, εξοπλισμό και μηχανήματα σαν και αυτά που χρησιμοποιούν τώρα, αλλά που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Και αυτό θα βοηθήσει και την βιομηχανία βέβαια, διότι για να τα παράγει θα έχει καταναλώσει λιγότερη ενέργεια. Ερχόμαστε σε επαφή και με τις οργανώσεις των καταναλωτών, αλλά και με μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους που μας υποστηρίζουν, διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε την Ευρώπη για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα. Το επόμενο θέμα, το επόμενο σημείο αφορά το πακέτο για τα απόβλητα και τα λοιπάσματα. Από την αρχή του κύκλου ζωής των προϊόντων μέχρι το τέλος, η... το πακέτο, το νομοθετικό πακέτο για τα απόβλητα είναι ένα κεντρικό σημείο, ένα κεντρικό στοιχείο για την κυκλική οικονομία και θέλουμε προφανώς ε, την γενική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την νομοθεσία για τα απόβλητα. Ο σημαντικός, ο εντυπωσιακός αριθμός των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί επαναεπιβεβαιώνει την προτεραιότητα που εσείς αποδίδετε ε, σε αυτές τις προτάσεις. Από ό,τι είδαμε από τις ε, συζητήσεις που έγιναν ε, για τις τροπολογίες το Σεπτέμβριο, υπάρχει μια ευρύτερη υποστήριξη και συμφωνία με την Κομισιόν σε πολλά θέματα, όπως είναι οι φιλόδοξες διατάξεις όσον αφορά την ξεχωριστή ε, διαλογή, των, την διαλογή των σκουπιδιών ή την πρόληψη αποβλήτων ή την ανακύκλωση. Ε, περιμένουμε να δούμε πώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή που από ό,τι καταλάβαμε θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο η προτινόμενη, ο προτινόμενος κανονισμός για τα προϊόντα των λιπάσματων είναι η πρώτη, λιπασμάτων, συγγνώμη, η πρώτη πρόταση που υιοθετήθηκε μέσα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και έχει σαν βασικό στόχο να ανοίξει την ε, ενιαία αγορά για ε, ανακυκλούμενα ε, λιπάσματα. Αυτός, αυτό περιμένουμε να οδηγήσει σε μια υποκατάσταση ή αντικατάσταση των ε, φωσφορικών ε, πρώτων υλών και με τον τρόπο αυτό να περιορίσουμε τις ε, ουσίες που μολύνουν το, το περιβάλλον. Η Κομισιό εξετάζει επίσης πώς μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε την αφαίρεση του καδμίου, την αφαίρεση του καδμίου μέσω οικονομικών ε, εργαλείων που έχουμε στην ε, διάθεσή μας, όπως το ΕΦΣΙ ή το Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη. Τώρα, οι σχετικές, όλες αυτές οι επενδύσεις, ε, δηλαδή το, σχέδιο, ε, το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη ή το ΕΦΣΙ αντιπροσωπεύουν μια πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα για την πράσινη οικονομία και ε, αποτελούν μια συγκεκριμένη συνεισφορά για να μπορέσουμε να αντλήσουμε και δημόσια και ιδιωτικά, και δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για τις πράσινες επενδύσεις. Ε, ας δούμε τι μπορούμε, ποια είναι τα κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ΕΦΣΙ υποστηρίζει μια σειρά project που αφορούν το περιβάλλον και την, αποτελεσματικότητα των, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, όπως το χάρη το project για το ανακυκλούμενο χαρτί ή το Novamont που είναι ένα χημικό project που αφορά ανανεώσιμες χημικές ουσίες στην Ιταλία. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε βέβαια ε, περισσότερο τον αριθμό των περιβαλλοντικών project που χρηματοδοτεί το ΕΦΣΙ, κυρίως ε, αυτά τα project τα οποία σχετίζονται με την κυκλική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΦΣΙ είχε μεγάλη επιτυχία την πρώτη χρονιά, η Κομισιόν πρότεινε το Σεπτέμβριο να παρατείνει την διάρκεια του ΕΦΣΙ μέχρι το τέλος του 2020 ανεβάζοντας ε, την, ε, τον στόχο για τις συνολικές επενδύσεις ε, σε τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ε, τους στόχους δε της Συμφωνίας του Παρισιού, η Κομισιό έχει προτείνει ότι τουλάχιστον το 40% των project ε, στην υποδομή του, του και στην, ε, και όσον αφορά την καινοτομία, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην κλιματική δράση σε συμφωνία με σκόπο 21 η ΕΕΦΣΗ αλλά επίσης ε, και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και ε, ταμεία και το τα, ταμεία επενδύσεων θα εξετάσουν θα εξετάσουμε το κατά πόσον μπορούμε να επενδύσουμε σε βιώσιμες και κυκλικές λύσεις. Θέλουμε βέβαια ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να προωθήσουμε τη γενικότερη οικονομία και να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια. Έχουμε επίσης Έχουμε δύο βασικά πρότυπα για την περιβαλλοντική ε, πολιτική. Ε, Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής ε, καταρχάς. Ούτως ή άλλως ε, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την, ε, το σχέδιο δράσης της κυκλικής οικονομίας. Όπως σας είπα, το 2017 θα σας παρουσιάσουμε ένα, μια έκθεση εφαρμογής, αλλά τέλος πάντων θα προχωρήσουμε με πέντε κυρίως πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι μια στρατηγική ε, για την καινοτομία που θα αφορά τα πλαστικά, ε, την χρήση και ε, την, επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των πλαστικών. Δεύτερον, ε, μια νομοθετική πρόταση για την ε, επαναχρησιμοποίηση του νερού. Θα ορίζουμε ελάχιστα ποιοτικά standards για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, αυτό τον πολύτιμο πόρο. Τρίτον, θα καλύψουμε το κενό στην, στο σύστημα ε, προμήθειας ε, νερού και θα υποβάλουμε μια αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Τέταρτον, θα κάνουμε μια, ένα κατάλογο πρωτοβουλειών που θα αφορούν ε, κάποια προϊόντα όπως τα χημικά και τα απόβλητα και εν κατακλείδη θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ελέγχου για να μετρήσουμε την πρόοδο της Ευρωπαϊ... που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την επίτευξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ας ξεκινήσουμε τώρα τον ε, πρώτο γύρο μιλητών. Από πλευράς ε, συντονιστών να δώσουμε το λόγο. Καλώ Καλό τους συντονιστές να σταθούν ε, στα δύο λεπτά έκαστος, γιατί έχουμε ένα κατάλογο μιλητών με 30 ονόματα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω με χαρά. Κύριε Αντιπρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και στην ακρόασή σας είχατε δεσμευτεί και θα ήταν πολύ χρήσιμο να το τηρείτε και όλα. Ευχαριστώ πολύ. Eco Design. Πριν από 10 χρόνια ήμουν από τους εμπνευστέ. Μετά στράβωσαν τα πράγματα με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και διάφορα άλλα θυμάστε. Ελπίζω και βλέπω και χαίρομαι ότι άλλαξε η οπτική γι' αυτό τώρα. Συνεισφέρατε κι εσείς ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Ποια κριτήρια ορίζεται λοιπόν για τους έξι παράγοντες ή τα προϊόντα αυτά που μας αναφέρετε και σε ό,τι αφορά τους πόρους ε, είναι αποδοτική, το απαντήσατε. Επιτέλους καταλαβαίνουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον ότι η περιβαλλοντική πολιτική δεν συνίσταται σε τιμωρίες και πρόστιμα αλλά σε επιστημονικά στοιχεία στην αρχή της παραγωγής έτσι ώστε το τελικό απόβλητο που δεν ανακυκλώνεται να είναι ε, όσο γίνεται λιγότερο. Δεύτερον, ένα παλιό μου έτσι, μέλημα και πόνος είναι πώς εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία. Κύριε Επίτροπε, να σας απαριθμίσω ε, πόσες ε, ρυθμίσεις εμείς έχουμε περάσει εδώ σχεδόν ομόφωνα και ε, ποια είναι η μοίρα του στα κράτη-μέλη και στη Γερμανία, τότε θα <laughs> σας πικράνω τόσο πολύ που και στο πρωινό θα σας φαίνονται πικρά αυτά που τρώτε το πρωί. Λοιπόν, παρακαλώ κλείστε τα αυτιά σας τις ειρήνες και να εφαρμόζονται αυτά σωστά. Για την κυκλική οικονομία έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Ε, όταν τέμνεται ε, το απόβλητο με τη χημεία, με τα χημικά προϊόντα. Το κατάλαβε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπονεί ένα νέο έγγραφο πλέον. Πόσο έχει προχωρήσει αυτό, μπορούμε να το εντάξουμε και να το συμπεριλάβουμε και στην κυκλική οικονομία. Γιατί η ανακύκλωση γίνεται όπως θέλεις, αλλά τελικά αν δεν ξέρεις ε, τι περιέχει το πλαστικό ή το, το τελικό απόβλητο, Πόσα λεπτά έχω ακόμα. έχω φάει το χρόνο μου. Ε, γιατί μετά θα πηγαίνουν για καταστροφή αυτά τα προϊόντα και δεν θα μπορούν να ανακυκλώνονται επειδή θα είναι επικίνδυνα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν για την παρουσία σας εδώ. Τρία κύρια ζητήματα. Πρώτον, ένα εισαγωγικό σχόλιο ειλικρινά μετά την αρχική απόσυρση του προσχεδίου πρόταση τη Επιτροπή για την Κυκλική Οικονομία που είχατε, είχατε υποβάλει ένα νέο ε, πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ένα σχέδιο δράση. Εμεί ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί γιατί δυστυχώ ε, θεωρούσαμε ότι κακώ δεν είχε ε, ενταχθεί σε μια νομοθετική πρόταση, γιατί δεν θέλουμε απλώ να αναφέρουμε την κυκλική οικονομία ως έναν ευσεβή πόθο που ποτέ όμω δεν ολοποιείται. Αναφερθήκατε στα έξι προϊόντα που ε, εσείς επιλέγετε για τον οικολογικό σχεδιασμό και λέτε ότι βασίζονται στις ενεργειακές τους ιδιότητες. Είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τη δέσμευσή της για τον οικολογικό σχεδιασμό, όμως θεωρούμε ότι το eco-design και αυτή η σχετική νομοθεσία είναι θεμελιώδης σημασία ε, για την κυκλική οικονομία. Όμως πρέπει να δούμε ε, τι μορφή θα λάβουν τα μελλοντικά προϊόντα, όμως πρέπει να μας πείτε κι εσείς κατά πόσο είστε πεπισμένος ότι θα υπάρχει σαφήνεια για τα υλικά που ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τα εφιστάμενα ε, προϊόντα και αγαθά, χωρίς ε, να καταφεύγουμε και πάλι στην εξόριξη πρώτων υλών. Ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι τα πλαστικά. Εδώ το σχέδιο δράση εντοπίζει δύο βήματα, με μια νέα στρατηγική για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία 2017 και εισαγωγή συγκεκριμένων δράσεων για την ε, μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων ε, στο πλαίσιο των ε, βιώσιμων στόχων ανάπτυξη του 2030. Θα ήθελα λοιπόν μια ενημέρωση από εσά για αυτέ τι δύο ενέργειε και κατά πόσο η Επιτροπή έχει αρχίσει να επεξεργάζεται αυτή την στρατηγική για το πλαστικό εντός του 2017 και κατά πόσο υπάρχει σχέδιο δράσης ε, από την Επιτροπή για τα κράτη-μέλη για να ε, περιορίσουν τα θαλάσσια απορρίμματα και πώς θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη Κομισιόν για την ε, ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Και το αναφέρω γιατί τελικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να μεριμνήσουμε ότι θα κάνουν τα δέοντα και θα υλοποιήσουν στο έπακρον τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κάτι τελευταίο, σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, υπάρχουν ορισμένες θετικές ε, πρωτοβουλίες από τον κλάδο και από τις ε, ΜΚΟ. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τα μέτρα ε, ακριβώς για τα πλαστικά απορρίμματα και το θαλάσσιο περιβάλλον στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής αυτής και το αργότερο όλα αυτά να γίνουν από το 2017. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάκρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κατάιναν, καλώς ήρθατε. Ε, μιλώ Ολλανδικά, την τρική μου. Κύριε Επίτροπε, είχα ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα ω ασχιώδη συζητητή εκ ονόματο των ε, Ευρωπαίων Στριπτικών Μεταρρυθμιστών για την ε, κυκλική οικονομία. Πρώτον, για την καινοτομία που αποτελεί προτεραιότητα στο σχέδιο δράση. Το λεγόμενο Innovation Deals είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά για να αποφύγουμε και να εντοπίσουμε τυχόν προσκόμματα, νομοθετικά προσκόμματα στο μέλλον ως προς την καινοτομία. Ε, Γιατί είναι είμαι απολύτως υπέρμαχος της σύστασης ε, δοκιμαστικών ε, πιλωτικών προγραμμάτων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη κάποια κράτη-μέλη, όπως το North Sea Research Roundabout, το οποίο ξεκίνησε φέτος και η χώρα μου, η ε, Φλάνδρα, αυτή τη στιγμή ε, συμμετέχει. Μετά, αυτά τα ευρωπαϊκά ε, πιλωτικά προγράμματα θα μπορούσαν να συσταθούν συμπληρωματικά. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα οικοδομικά απορρίμματα, ε, υπάρχει αυτό το recycling protocol το οποίο έχει ανακοινωθεί για το 2017. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γι' αυτό και ποια είναι η σύνδεσή του με τους υποχρεωτικούς στόχους σε ό,τι αφορά αυτά τα απορρίμματα για το 2020 στο ε, πλαίσιο για τα πόδια. Ε, για τα και τα βάζα. Ε, μέχρι το 2025 και μέχρι το 2030 τι θα γίνει αντίστοιχα. Και το και ευρύτερο ερώτημα προς τον Επίτροπο, το σχέδιο δράση συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες ε, για την ε, παροχή κινήτρων για τα δευτερογενή απορρίμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε πλήρως. Όμω, αντίστοιχα πρέπει να ε, δώσουμε κίνητρα και για τον περιορισμό, την αποφυγή, αν θέλετε, της ε, δημιουργίας ε, απορριμμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία πλήρη ε, πολιτική και σωστά επεξεργασμένη, ούτω ώστε να κρατούμε υπό έλεγχο αν θέλετε, την δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβετε υπόψη, θεωρώ, κύριε Επιτροπέ. Και κάτι τελευταίο είναι σημαντικό να το αναφέρουμε γιατί ήμουν εισηγητή και για την ε, έκθεση για την βιοπικιλότητα που πρόσφατα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσατε να μα πείτε αν υπάρχουν νέα σε ό,τι αφορά το fitness check για τι οδηγίε ε, για ε, του βιοτόπου και θεωρείτε ότι λειτουργούν και ότι εφαρμόζονται πλήρω. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερμπράντη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Κατάινεν που ήρθατε. Πρέπει να αρχίσω λέγοντας ότι αισθάνομαι κάπως παγιδευμένος μέσα σε ένα τέτοιο κύκλο και δεν συνδέεται αυτό με την κυκλική οικονομία. Κάθε έξι μήνες καλούμε τον Αντιπρόεδρο να μας πει τι γίνεται και ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την κυκλική οικονομία και τα αντίστοιχα μέτρα της δέσμες, γιατί δεν ήμασταν πάρα πολύ βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφήρμοζε αυτά που υποσχέθηκε ότι θα έκανε. Αλλά τώρα αισθάνομαι ότι προσπαθεί ο Επίτροπος να μας πείσει για όλα αυτά τα ωραία και τα θαυμαστά της κυκλικής οικονομίας. Μα γι' αυτό σας καλούμε εδώ κάθε εξάμεινο. Εμείς είμαστε ε, ακρεφνείς υποστηρικτές της κυκλικής οικονομίας και θεωρούμε ότι είναι ουσιώδης μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξακολουθούμε να πιέζουμε και δεν χαλαρώνουμε τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνετε περισσότερα από ό,τι κάνετε. Και είναι και απαραίτητο. Αν δω ε, το πρόγραμμα δράσης και όλες τις διαφορετικές δράσεις, σχεδόν όλες έχουν καθυστερήσει, σχεδόν όλες υποθέτω ότι είναι τυχαίο τελείως σύμπτωση. Ε, σήμερα τη μέρα που είστε εδώ και πάλι ε, κάνετε μια ανακοίνωση μαζί με την ΔΕΙΟ για ε, τον οικολογικό σχεδιασμό. Ελπίζω σε έξι μήνες από τώρα να μας κάνετε νέες εξαγγελίες αλλά να μας μιλάτε για υλοποιημένα μέτρα και θα χαρούμε πολύ γι' αυτό. Επίσης χάρηκα με τα σχόλια σας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ε, ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τα μεγάλα πράγματα και τα σπουδαία πράγματα και αυτό είναι η κυκλική οικονομία. Και ο Φραντ Τίμερμανς, ο συνάδελφός σας, τα λέει αυτά, αλλά ο κύριος Γιούγκερ συνδηγεί ηχθείως και ε, παρακολουθώ πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη και έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Ιούνκερ και το επιτελείο του εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτά είναι κάτι μικροπράγματα που δεν θα πρέπει να ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζω και στον Economist ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τον ίδιο λαϊκισμό ε, για τον οποίο κατηγορεί κάποιου άλλους ε, μη προτείνοντας αυτά που θα πρέπει και για τις τοστιέρες και για τους καταλήτες και ξέρετε για τι πράγματα μιλάω. Ε, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανισχύει λιγότερο για το βρετανικό λαϊκό τύπο και περισσότερο για τη δική μας οικονομία. Τι χρειάζεται, αλλαγή νοοτροπίας, όχι ωραία λόγια, αλλά και πολύ ισχυρή δράση και όχι ε, μεσοβέζικα πράγματα που ακούμε τώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι λέει η δέσμη για τον οικολογικό σχεδιασμό. Θα δείξει. Ένα τελευταίο παράδειγμα και θα τελειώσω τις ερωτήσεις μου, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα της απόδοσης ε, των πόρων ε, υποτίθεται ότι θα ήταν μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα έχει βγει. Προτίθεστε να το ξαναβάλετε γιατί αν θεωρούμε ότι είναι σπουδαίο και μεγάλο πράγμα, πολύ σημαντική μετάβαση της οικονομίας, εκεί είναι η θέση της. Και πολύ τελευταία ερώτηση για το οικολογικό σχεδιασμό. Μόνο στην ενέργεια εστιάζεται ή και στη χρήση των πόρων, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της επόμενης φάσης του οικολογικού σχεδιασμού. Ευχαριστώ. Very much, Miss Ευχαριστώ κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω τις ερωτήσει. ερωτήσεις. Ε, και εγώ χαίρομαι, όπω και άλλοι συνάδελφοι, που είπατε ότι ο οικολογικό σχεδιασμό ε, είναι ε, μεγίστη σημασίας, όμως περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό να δούμε κάτι αυτό. Μας έχετε υποσχεθεί το πρόγραμμα αυτό από την αρχή τη θητεία μα και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια οδηγία που θα μπορούσε να επιλύσει πολλά ζητήματα που αφορούν την κυκλική οικονομία αλλά και γενικότερα την διαχείριση απορριμμάτων. Περιμένουμε λοιπόν και θα θέλαμε να δούμε κάποια βελτίωση. Θα θέλαμε να μας ε, δώσετε, να μας παρουσιάσετε ρεαλιστικά τις ε, προοπτικές και πώς ε, μπορεί να αποδοθεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε διάφορες πρωτοβουλίες στην ομιλία σας. Όμω, αναφερθήκατε μόνο επιγραμματικά σε αυτές. Θα θέλαμε να μην τι κατονομάζετε μόνο, αλλά να μας ε, μιλάτε, να μας παρουσιάζετε το περιεχόμενό τους, ε, την διασύνδεσή του, με την γενικότερη έννοια της κυκλικής οικονομίας. Και το τρίτο μου ερώτημα αφορά την ε, κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με αυτά τα απορρίμματα και υποβλητά προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε αρνητική διάκριση εναντί της ε, ενεργειακής κατανάλωσης ε, των απορριμμάτων. Ό,τι απομένει λοιπόν ως απόρριμα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται και όχι να καταλήγει στη χωματερή. Και οι μελλοντικές γενιές ενδεχομένως να έχουν ε, μια καλύτερη κατάσταση στα χέρια τους. Επομένω, ε, νέα χρήση των απορριμμάτων και όχι χωματερές. Ευχαριστώ κύριο Σάικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ξέρετε ότι το σχέδιο δράσης έχει ορίζοντα ενός έτους ή μάλλον εδώ και ένα χρόνο το έχουμε στη θέση μας, ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο. Αν δείτε τι έχει γίνει με το σχέδιο δράση τώρα, βέβαια, είναι λίγο απογοητευτικά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση ε, για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μετά από ένα χρόνο, κατά τα λοιπά, και συναδελφοί μου θα έχουν κάποια ερωτήματα και άλλα ζητήματα που βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει και τίποτα αυτό. Τουλάχιστον δεν το έχουμε δει εμεί. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν σχεδίου δράση, δεν είναι και πολύ θετικό το αποτέλεσμα έω τώρα. Α εστιάσουμε όμω την προσοχή μα στον οικολογικό σχεδιασμό. Αναφερθήκατε στα 6 στοιχεία που υπάρχουν στον κατάλογο. Αρχικά είχαμε 12 όμω. Έξι φύγαν λοιπόν. Πρέπει να υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι για να γίνει αυτό, γιατί ε, επαναλαμβάνω αυτό που είπατε κι εσείς, ε, ότι με τον οικολογικό σχεδιασμό έχουμε κατανάλωση χαμηλότερης ενέργειας που είναι φτηνότερη για αυτό και στους καταναλωτές, χαμηλότερες εισαγωγές. Καλό αυτό λοιπόν για την ενεργειακή μας εξάρτηση ιδίω από την Ανατολή. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία γίνεται πιο ανταγωνιστική, γιατί συνήθως είναι καλύτερη η δική μας βιομηχανία στις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Είναι καλύτερο για το περιβάλλον όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Το μοναδικό πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι το διάσημο και εξαιρετικά γνωστό ε, νομοθετικό άχθος. Πάντα το επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσο επαχθές είναι πια το να πηγαίνει κανείς σε ένα κατάστημα και να μπορεί να βρίσκει μόνο την ενεργειακά αποδοτική συσκευή και όχι την άλλη την παλιά. Τι σας ε, δημιουργεί πρόβλημα. Τίποτα. Μόνο οι βρετανικέ κίτρινες βλάδες είναι αυτέ που λένε ότι θα χαθούν πια ε, τα αγγλικά ε, προγεύματα. Και εσεί του ακούτε, γιατί έτσι φεύγουν ε, οι συσκευέ. οι φρυγανιέρε. Ενώ για παράδειγμα στον κατάλογο έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που τα έχετε, ενώ άλλα τα έχετε βγάλει χωρίς κανένα άλλο λόγο. Επομένω, απλά φοβάστε τις Βρετανικές φυλάδες. Αυτή είναι η ουσία. Για ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, το θεωρώ πολύ μεγάλο κρίμα, ε, που βάζετε ένα τέλος σε αυτό το θέμα ως Κομισιόν. Ο οικολογικός σχεδιασμός τώρα είναι το πρώτο στοιχείο που ε, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ε, σχεδίου δράσης και δεν είναι μια πολύ καλή αρχή. Σας ευχαριστώ κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα λόγια σας και ελπίζω ότι όλες αυτοί οι ευσεβείς πόθοι δεν θα μείνουν ευσεβείς πόθοι ε, μέσα σε αυτή που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα, αλλά θα αποτελέσουν ε, την βάση για την υλοποίηση μιας πραγματικής ε, κυκλικής οικονομίας. Μιλήσατε για τις προθεσμίες και αναφερθήκατε κυρίως στα πλαστικά τα οποία καταλήγουν είτε στην φύση είτε στη θάλασσα. Δεν είπατε όμως τίποτα για αυτό το απαραίτητο στάδιο το οποίο πρέπει να υπάρχει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή όλες οι άμεσες ή έμεσες επιδοτήσεις όσον αφορά τα, ο, τα ορυκτά καύσιμα. Ξέρω ότι βέβαια μιλάμε για, ε, υπάρχει επίτροπος ενέργειας και πετρελαίου προφανώς. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε υιοθετήσει ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητάμε την κατάρκηση όλων των επιδοτήσεων όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα τι θα πιστέψουν οι πολίτες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη της ε, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελούν την, ε, ε, την έκφραση της θέλησης των πολιτών. Θέλουμε, θέλει η Κομισιό να ικανοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών ή να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας ε, υιοθετείται κυρίως από το πακέτο για τα απόβλητα και η εφαρμογή αυτών των τεσσάρων οδηγιών ε, και τα όσα έχουμε κάνει δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Όμως έχουμε 1.700-1.700 τροπολογίες στις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτό δείχνει πώς εφαρμόζεται αυτή η κυκλική οικονομία. Και ναι, μεν μπορεί ο δρόμος να είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις, όμως ο δρόμος αυτός δεν οδηγεί στην σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση, η, η εκθέσεις αυτές ε, έχουν ε, ε, προκαλέσει αντιδράσεις από τα κοινοβούλια της Γαλλίας και της Αυστρίας. Υπάρχουν πολλά, πολλές αμφιβολίες για την κυκλική οικονομία, διότι θεωρούμε, όχι για την ίδια την κυκλική οικονομία, αλλά για τις προτάσεις που, κάνουν, που κάνει η Κομισιόν, που θεωρούν ε, πολλοί ότι έχουν σαν στόχο μόνο την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Ε, πιστεύουμε ότι μπορούν να υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει μια ουσιαστική κυκλική οικονομία, πολλές ε, ε, πολλά δημοσιεύματα στον τύπο μας πείθουν ότι γίνεται αυτό. Βέβαια στηρίζεται περισσότερο τα όσα γίνονται ε, στην πρωτοβουλία των πολιτών. Ξέρουμε πολλά παραδείγματα ε, εταιριών και επιχειρήσεων που έχουν εσωτερικεύσει την ανακύκλωση των ε, προϊόντων τους και όλα βέβαια γίνονται σε κλίμακα κάθε εταιρεία. Υπάρχει επομένως αυτή η ευελιξία σε ε, επίπεδο επιμέρους ε, επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε όμως να το γενικεύσουμε. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω, να, ε, να μας πείτε δηλαδή τι γίνεται, τι, πιστε, τι θα πρόκειται να κάνει η Κομισιό. Επίσης η παλαιότητα είναι ένα θέμα που αφορά την κυκλική οικονομία, ενώ Ταυτόχρονα εμείς εισάγουμε από την Ανατολική Ασία προϊόντα τα οποία μπορούν να κατηγορηθούν για τέτοιου είδους, ε, για παλαιότητα τέλος πάντων, ε, το ότι είναι φθαρμένα. Θα πρέπει να, θα, δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, μεταφορά των ε, βιομηχανιών μας, ε, των επιχειρήσεών μας και θέλει να μου πει και η Κομισιόν πώς ε, μπορεί να αντιμετωπίσει την προγραμματισμένη παλαιότητα των προϊόντων μας. Ευχαριστώ. Εδώ είχαμε την πρώτη ενότητα ερωτήσεων. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κατάινεν για να απαντήσει. Έτσι συνολικά. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι όσα έχουμε κάνει είναι άχρηστα, είναι πολύ αργά, είναι πολύ λίγα και μαύρα χάλια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή αρχή. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία θέλουμε να καταφέρει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρώτη νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή θα ήταν μια καλή αρχή για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία. Μη, μη. Λέω, το είπα, θα σας προβοκάρω, γιατί με προβοκάρετε κι εσείς και με προκαλείτε. Λοιπόν, ε, νομοθετική πρόταση για τα απόβλητα. Εγώ κατάλαβα ότι το Γενάρη θα το ψηφίσετε. Γιατί το Γενάρη, γιατί έχει το Δεκέμβρη Υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος. Όσο το γρηγορότερο, τόσο το καλύτερο. Γιατί να περιμένουμε μέχρι τον Γενάρη. Τι άλλο. Για ε, τον κανονισμό για τα λοιπάσματα. Έχει φτάσει ήδη. Μήνες ολόκληρος τώρα περιμένει. Δεν χρειάστηκε για μας τόσο πολύ καιρό για να προτείνουμε την νομοθεσία. Όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Κατανοώ ότι πολιτικά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξετε σε συμβιβασμούς για τα θέματα αυτά. Αλλά ας μην επικρίνουμε τα θετικά. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος όταν έχουμε κοινό στόχο. Επίσης, αν απλώ επικρίνουμε την οδηγία για τον οικολογικό συνδυασμό, η νέα πρόταση που πάει τώρα στην Επιτροπολογία, αυτό βοηθάει εκείνου που είναι βασικά πολέμοι τη οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Κάποιοι θέλουν λιγότερα, κάποιοι θέλουν περισσότερα, αλλά τελικά έχουμε ένα κατάλογο έξι ειδών ε, που έχουν επιλεγεί γιατί είναι από τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης συνέργειας. Και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν τερματίζει εδώ. Καλό θα ήταν λοιπόν να βρούμε λίγο πιο θετικό έδαφος για να συνεννοηθούμε για την κυκλική οικονομία. Ξέρω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να κριτικάρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα στραβά ψωμιά εμείς τα κάνουμε. Αλλά θα πρέπει τα καλά να τα προβάλλουμε στους πολίτες. 99,99% των πολιτών δεν καταλαβαίνουν τι εστί κυκλική οικονομία. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προβάλλουμε αυτή την ιδέα στους πολίτες. Ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή... Ε, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο και θα παραμείνει ηγέτη και στο μέλλον, αλλά εμεί ε, ω ρυθμιστέ, ω νομοθέτες θα πρέπει να πούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην γραμμική και την κυκλική οικονομία και να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ λύσει. Η εφαρμογή και η υλοποίηση παραμένει πρόβλημα και για το μέλλον. Ιδιαίτερα για τομεί πολιτική που είναι καλά ανεπτυγμένοι. Υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής. Του χρόνου το 2017 θα ενταθούν οι προσπάθειες υλοποίησης με τρεις πρωτοβουλίες για τη συμμόρφωση, για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αναφορά. Ε, χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποδώσει. Υπάρχουν κανόνες, θα πρέπει να εφαρμόζονται και σωστά. Κοιτάξτε, θα πρέπει να παρακολουθούμε τα κράτη-μέλη ε, στη συνειδητοποίηση της νομοθεσίας σε όλα τα θέματα, όχι μόνο για την κυκλική οικονομία και για την έννοια αγορά. Για τη στρατηγική για τα πλαστικά δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, διότι τώρα μόνο ξεκινάει αυτή η δουλειά και θέλουμε να συμπεριλάβουμε ε, όσο γίνεται περισσότερους ενδιαφερομένους. Κυρία Ντάλη, εσείς αναφερθήκατε σε αυτό και πολλούς από τους κρίσιμους τομείς που θα πρέπει να ε, λύσουμε. Εύκολο δεν θα είναι, αλλά είμαι βέβαιος ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση και υπάρχει θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Η στρατηγική λοιπόν για τα πλαστικά ελπίζουμε να βελτιώσει και τις επιδόσεις και τις αποδόσεις ε, με την καινοτομία, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Ε, ελπίδα μας είναι να αντιμετωπίσουμε ε, τρία πράγματα με τη μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά, την χαμηλή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πλαστικών και ε, την ρήπανση στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο και στους ωκεανούς. Η θαλάσσια ρήπανση από πλαστικά είναι ένα θέμα ε, που αναδύεται τώρα και κερδίζει έδαφος στην προσοχή της κοινή γνώμης παγκοσμίω. Ελπίζουμε και περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα μέχρι τα τέλη του 2017. δηλαδή το φθινόπωρο ή το χειμώνα, γιατί χρειάζεται χρόνο να καταρτιστεί αυτή η πρόταση. Για την καινοτομία βεβαίως και τις συμφωνίες για την καινοτομία, πώς έχει η κατάσταση. Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος έκλεισε στις 15 Σεπτεμβρίου, 32 δήλωσαν ενδιαφέρον από διάφορα κράτη-μέλη, 14 τον αριθμό. Είναι καινούργια τελείω διαδικασία αυτή. Είναι θέματα που αναφέρονται ε, στις αιτήσει ποικίλουν από θέματα που έχουν να κάνουν για το ε, είδωρ, τη συνεργατική οικονομία και καινοτομίε σε διάφορους κλάδους. Τώρα επιλέγουμε τα πρώτα έργα. Τον Νοέμβριο θα ενημερώσουμε τους ετούντες, πολύ σύντομα δηλαδή, Πέντε επιλέγονται. Θα ανακοινώσουμε ποια είναι αυτά τα πέντε έργα και θα υπάρξει μια κοινή δήλωση για να αρχίσει αμέσως ε, μετά η ε, ουσιαστική δουλειά. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες και η νέα αγορά τους. Είναι μια από τις μεγαλύτερες διορθωτικές αλλαγές που μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη, ακριβώς για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε διάφορους τομείς. Και θα πρέπει να δούμε κάθε τομέα από άλλη σκοπιά. Ας πούμε, τα πλαστικά χρειάζονται δική τους ρύθμιση. Ε, άλλα δευτερογενή προ, ε, πρώτες ύλες, άλλα υλικά χρειάζονται άλλη νομοθεσία. Εδώ λοιπόν θέλει πολύ δουλειά, όχι μόνο για τον χρόνο, αλλά και για τα επόμενα έτη. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία αγορά εσωτερική με ένα κανόνα για όλα τα υλικά για όλες τις ύλες αυτές, Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία αγορά εμποδίζει και τις επενδύσεις και τη λειτουργία της κυκλικής οικονομίας και εργαζόμαστε στο θέμα αυτό. Ενεργειακή απόδοση κατά πόσο θα πρέπει να εντάσσεται στο ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν θυμάμαι πρέπει να σας πω αν το αναφέραμε την περασμένη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να δίνουν έμφαση εκεί όχι μόνο στα κτίρια, αλλά και στην υπόλοιπη νομοθεσία που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Διακόπτει ο κύριος Γερμπράντη. Ναι. Ε, και αποδοτικότητα των πόρων. Α, ναι, άλλο αποδοτικότητα των πόρων και άλλο ενεργειακή απόδοση. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Διότι πώς αξιολογείται αυτό, πώς εκτιμάται. δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Δεν είναι εύκολο να μετρηθεί αυτό. Γιατί δεν υπάρχει και σαφής ορισμός για το πώς υπολογίζεις την απόδοση των πόρων. Και πώς υπολογίζεται αυτό αναλόγως αν ε, εισάγονται ή εξάγονται από τη μία χώρα στην άλλη η πόροι αυτοί η φυσικη Και έρχομαι στην ε, οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και το μέλλον της. Εάν οδηγία αυτή ε, με τη σημερινή μορφή της θεωρείται βελτιωμένη, αποτελεί βελτίωση για την ενεργειακή απόθεση. Το να αλλάξει, να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία ε, του ε, οικολογικού σχεδιασμού δεν είναι τόσο προφανές και εύκολο. Θα πρέπει να, να δούμε κάποια στοιχεία όπως είναι η διάρκεια, η ε, δυνατότητα επισκευής και χρήσης. δηλαδή είναι θέματα περίπλοκα. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο τώρα φυσικά για να επεκταθεί η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Γιατί επικρατεί εντύπωση που είναι πάρα πολύ αρνητική. Πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. The, uh, και ελπίζουμε να το, να το διευρύνουμε και να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Αναφέρω το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΨΙ. Και επενδύσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Ιδιαίτερα ε, έργα για την κυκλική οικονομία, παρόλο που σας ανέφερα λίγα, παραμένουν πολύ λίγα για μένα. Για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, πολλές επενδύσεις στην κυκλική οικονομία είναι τόσο επικερδείς που μπορούν να βρουν κονδύλια από την αγορά, ελπίζω, και η άλλη εξήγηση μπορεί να είναι ότι οι επενδυτές της κυκλικής οικονομίας δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει το ΕΨΙ, Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, και δεν ε, υποβάλλουν αιτήσει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι το λεγόμενο blending, ε, ο συνδυασμός των διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΦΣΥ, ιδιαίτερα στη διαχείριση αποβλήτων. 6 δισεκατομμύρια ευρώ περιμένουν από τα διαρθρωτικά ταμεία να βελτιώσουν ε, τη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο για να πιάσουν τόπο. Όχι απλώς να αντικατασταθούν οι παράνομες χωματερές από νόμιμους χιτά, αλλά να ανακυκλώνεται σωστά ε, ε, η ποσότητα αυτή των αποβλήτων και να επαναχρησιμοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν συνειδητοποίηση και αυτό μπορεί να το κάνει το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, να ε, πλαισιώσει και να συμπληρώσει το χρηματοδοτικό πακέτο από τα διευθυντικά ταμεία. Παρακαλώ να το διαδώσετε αυτό και στις εκλογικές σας περιφέρειες. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα. Αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και άλλο γύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τις πρώτες ε, απαντήσεις αυτές, έχουμε λάβει ορισμένα από μέλη ε, που θέλουν να δευτερολογήσουν και να σχολιάσουν τις απαντήσεις σας. Να επενθυμίσω μόνο για να κλείσει και αυτή η αψημαχία, ότι περιμένουμε μια πιο φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής εδώ και ένα χρόνο. Και νομίζω ότι είναι κοινή η ευθύνη και ενώπιον μιας ε, πολύ μεγάλης και περίπλοκης ε, πρότασης και εμείς εργαζόμαστε επί της πρότασης αυτής με πάνω από 2.000 ε, τροπολογίες που είναι δύσκολο να καταλήξει σε συμβιβασμό. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Καλό τα μέλη ε, να τηρούν το χρονικό του όριο. Η κυρία Γκβοστέτ έχει το λόγο. Ο κύριο Φλόρεν νομίζω ήθελε να πει κάτι, αλλά δεν πειράζει. σω θα πρέπει να το πει στο τέλο. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, σα ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μα συζητούμε για τα θετικά της κυκλικής οικονομία. Όμω, ε, θα ήθελα να μιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο κλάδο τον, ε, ε, του λάστιχου. Είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως και τρεις φορές και έτσι να γλιτώσουμε, να συγκονομήσουμε 5 κιλά ε, πρώτων υλών, κατά 20% να μειώσουμε τις εκπομπές και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτά τα προϊόντα βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα λάστιχα αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ασία και ακόμα και καινούργια όταν είναι, είναι πολύ λιγότερο ασφαλή και εξοικονομούν πολύ λιγότερη ενέργεια. Επομένω, πώ θα τα εντάξετε αυτά τα προϊόντα που είναι τόσο σημαντικά σε αυτόν τον κλάδο τη κυκλική οικονομία. Δεύτερον, μιλήσατε για τα θαλάσσια απόβλητα. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο στο σχέδιο δράση σα. Θέλετε να περιορίσετε τον ε, όγκο του, ε, όμω ε, θα ήθελα να μιλήσω και για συγκεκριμένα Συγκεκριμένε ουσίε ε, που εντάσσονται μεταξύ άλλων και στα καλλιτικά, γιατί αυτά ε, δεν μπορούν να τύχουν επεξεργασία ε, στα συστήματα και γι' αυτό απελευθερώνονται στου ωκεανού. Ποια θα είναι η στρατηγική σα, λοιπόν, πώ εντάσσεται όλο αυτό στο σχέδιο δράση σα, θα υπάρξει σχέδιο δράση απέναντι σε αυτέ τι επιχειρήσει που ε, καταναγκάζονται να βρουν εναλλακτικέ λύσει και θέλουν έτσι να εξαλείψουν τη χρήση αυτών των ουσιών. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Επιτρέψτε μου ορισμένε προτάσεις βελτίωσης. Ε, θα προσπαθήσω κι εγώ να μην είμαι επικριτικός, αλλά επικοδομητικός. Να σας κάνω προτάσεις βελτίωσης ω προ τα όσα μας προτείνετε. Πρώτον, για την ε, διατροφική σπατάλη, τη σπατάλη τροφίμων δηλαδή, στην οδηγία σας δεν υπάρχει στόχος για τον περιορισμό ε, της ε, σπατάλης τροφίμων. Πάνω από 100, εκατομμύρια τόνοι τροφίμων όμως ε, σπαταλώνται κάθε χρόνο και μπορούμε να φτάσουμε και στους 120 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Επομένως, τι θα γίνει ως προς αυτό, τον, ως προς αυτό το σημείο, όπως σε σχέση και με τα όσα είπε και η κυρία Μποναφέ, που θέλει να ε, περιορίσουμε τη σπατάλη μέχρι, κατά 50% μέχρι το 2030. Δεύτερον, η προγραμματισμένη εξάλληψη συγκεκριμένων συσκευών βλέπουμε ότι ο χρόνος ζωής ε, τα τελευταία χρόνια για τους υπολογιστές για παράδειγμα από τα 12 έτη ζωής το 1980 έχουμε περάσει τα 4 έτη πλέον. Επομένως, οι συσκευέ μα βλέπουμε ότι έχουν πολύ μικρότερο ε, χρόνο ζωή. Αυτό έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει ε, και στο περιβάλλον και οικονομικέ και κοινωνικέ ε, προεκτάσει. Πώ όλα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο δράση σα και θεωρείτε ότι θα υπάρχει κάτι ε, ως ανεξάρτητο εργαλείο μέχρι το 2020. Τρίτον, μιλήσατε για τον Όχ Παντεκαλέ που το 2014 στο master plan του είχε ε, προβλέψει 0% ε, εκπομπές διευθυντήτων του ανθρακά μέχρι το 2050. Μπορείτε να έρθετε να βρείτε τους νέους ε, ηθήνοντες αυτής της περιφέρειας, γιατί από μετά τις εκλογές του 2015 δεν ακούμε πια τίποτα. Τη γνωρίζω αυτή την περιφέρεια, γιατί αυτή είναι και η δική μου εκλογική περιφέρεια στα προεδρικά της Γαλλίας. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί το 2013 λοιπόν είχε ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επιχείρηση της ε, τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Η κυρία Γκέλεγγ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Θα ρώταγα για τα πλαστικά. Η Μίριαμ την έκανε όμως ήδη, άρα θα περάσω στη δεύτερη ερώτηση. Δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά θεωρώ ότι οι, απαντήσεις σας είναι ελιπέστατες. Γι' αυτό πρέπει να ξαναθέσω το θέμα των ε, πλαστικών, κυρίως ε, σε σχέση με το σχόλιο σας ε, ότι μας παίρνει πολύ χρόνο για να κινηθούμε. Μιλώντας για την κυκλική οικονομία, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα συμπεριλάβουμε τα πλαστικά, ότι πρέπει να περιμένουμε ε, τα πλαστικά που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το λιγότερο ανακυκλούμενο προϊόν. Πρέπει να περιμένουμε ένα άλλο έγγραφο της Κομισιόν. Είναι τρελό αυτό να μας λέτε ότι εμείς χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να κινηθούμε όταν περιμένουμε ε, μια πρόταση για τα πλαστικά. Κυρίως όπως είπε και η κυρία Γλώστα, το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε μια απόφαση Το μεγάλο θέμα είναι οι μικροϊνες που ε, προέρχονται από τα πλαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τα ενδύματα. Αυτό είναι το βασικό το μεγάλο πρόβλημα. Και μας είπατε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα πρόταση. Εγώ δεν κάνω συνήθως κριτική προς την Κομισιό, αλλά θεωρείτε ότι είναι σωστό να αρχίσετε να, λάτε, να μας μιλήσετε για την κυκλική οικονομία και να μας λέτε «Α, για τα πλαστικά δεν θέλω να μιλήσω». Ακόμα δεν το έχουμε ολοκληρώσει και δεν θέλω να πω τίποτα. Λοιπόν, ε, εμείς θέλουμε να ξέρουμε όμως τι, τι προτίθεστε να κάνετε. Ο κύριος Τόβας, δεν σας είχα δει, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω στη συνάντησή μας ε, τον κύριο κατάνι Κατάινεν. Αυτά στα φιλανδικά. Περνάω στα αγγλικά. Πώς ε, θα διατηρήσουμε μια ε, μοραλιστική ε, ε, ενιαία προσέγγιση στα διάφορα θέματα που αφορά την σπατάλη των τροφίμων, βιομάζα, υλικά, αντιμετώπιση αποβλήτων κτλ. κτλ. Γιατί έχω την εντύπωση πολλές φορές ότι προωθούμε κάποιες πολιτικές μόνο, ενώ θα έπρεπε όλες οι πολιτικές μας να ε, ταιριάζουν η μία με την άλλη, να οδηγούν προς έναν συγκεκριμένο στόχο. Λοιπόν, επίσης τεχνολογική ουδετερότητα, έστω και αν δεν έχουμε φτάσει σε κάποια ε, επίπεδα ε, αυτή τη στιγμή, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε λίγα χρόνια ε, με ένα σοβαρότατο πρόβλημα στα χέρια μας, κυρίως οι μικρές χώρες. Τρίτο είναι η αποτέφρωση. Η αποτέφρωση σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Να τι γίνεται στην Νάπολη και η Καμόρα πώς χρησιμοποιεί την αποτέφρωση μάλλον το αντιμετωπίζει με διαφορετικά τρόπο από ότι οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δούμε πολλές φορές τις διαφορές στα διάφορα είδη των αποτεφρώσεων και τις ε, οικονομικές συνέπειες. Και αυτό Ε, και αυτό είναι πολλές φορές εις βάρος της αποτέφρωσης. Αυτές ήταν οι σύντομες ερωτήσεις που ήθελα να σας θέσω. Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε Κατάινεν, θα ήθελα να ε, τονίσω ένα πρόβλημα που έχουμε που δεν έχει να κάνει μόνο με την κυκλική οικονομία αλλά κυρίως με την επισητιστική ασφάλεια. Μιλήσατε για 140 ή 150 δισεκατομμύρια που χάνει η Ένωση κάθε χρόνο από τη σπατάλη τροφίμων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ε, να βρει μια κοινή μεθοδολογία για την εναρμόνιση όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Θέλουμε να απευθύνουμε μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει. Γιατί βλέπετε ότι η γεωργία είναι από τις μεγαλύτερες πηγές ρήπανσης. Έχουμε και τη Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χάνεται πάρα πολύ ενέργεια ε, για να παράγουμε τόσα πολλά τρόφιμα που πετάμε μετά και παράγουμε και πολλά σκουπίδια. Το κόστος είναι πολλαπλάσιο από εκείνο που θα μπορούσαμε ε, να υπολογίσουμε από την ε, άμεση σπατάλη τροφίμων. Πολλά κράτη-μέλη ενδιαφέρονται πάρα πολύ να εργαστούν σε αυτό το τομέα και περιμένουν από τις Βρυξέλλες επιτέλους να κάνει μια κοινή πρόταση για να ορίσει μια κοινή μεθοδολογία για να έχουμε εναρμονισμένη ε, στάση απέναντι στο πρόβλημα και να το λύσουμε γρήγορα. Ερώτηση δεύτερη. Η ίδια η κυκλική οικονομία και το υπόδειγμα αυτό, δηλαδή ότι έχουμε δευτερογενείς πρώτες ύλες ε, από την ανακύκλωση. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά υλικά όμως που έχουν τοξικά στοιχεία και κατάλοιπα. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Υπάρχει το πρόγραμμα Horizon 2020 που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε Ας περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα νέα προϊόντα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αντιδράσει. Ε, ξεχνάμε λοιπόν ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μια πρόταση ε, για την ανακύκλωση για να μην πετάμε τόσο πολλά τρόφιμα. Ξέρουμε ε, ότι θέλουμε να προχωρήσουμε αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Ο ε, κύριο Φλόρενς, κύριε Κατά, κύριε Αντιπρόεδρε, για λόγου συναδελφικού θα πρέπει να μιλήσω για την κυρία Μποναφέ. Ε, κάνει ό,τι μπορεί ε, και μας πιέζει πάρα πολύ και βοηθή μου βλαστημάνε που δουλεύουν μερόνυχτα ολόκληρα και Σαββατοκύριακα. Δεν φταίει η συγγήτρια. Εξηγήστε σε ένα Βούλγαρο, ένα Ρουμάνο, είναι πολύ δύσκολο. Τι στόχους έχουμε. Και θα έρθετε να δείτε πώς θα ζητοκραβεγάσουν στη δική μου πολιτική ομάδα. Δεν πρόκειται να το ζήσετε αυτό τόσο γρήγορα. Καταλαβαίνω και τους νέους. Ο κύριος Ποτότσνικ έκανε μια καλή πρόταση και ο Γιούγκερ ε, σαν ήταν το λικός Γιούνκερ το ε, διεκπαιρέωσε σαν να μην υπήρχε. Γι' αυτό οι νέοι μας ε, εξοργίζονται και ανησυχούν. Ήταν καλή η πρόταση του Ποτότσνη, καλά. κύριε Επίτροπε, ο Επίτροπος Βέλα έχει ακόμα δουλειά να κάνει. Υπάρχουν ακόμα τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα ανοιχτά. Και δεν μπορεί να εγκριθεί αυτό όπως έχει από τους πολιτικούς. Θα πρέπει να πατήσει λίγο γκάζι ο κύριος Βέλα, ο συνάδελφός σας εκεί στην Επιτροπή, για να μας φέρει κάτι να το εγκρίνουμε. Ευχαριστώ κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κατάινεν, που ήρθε σήμερα εδώ μαζί σας. Προφανώς το, το πέρασμα από μια γραμμική οικονομία σε μια κυκλική οικονομία δεν είναι μια επιλογή, είναι μια υποχρέωση την οποία έχουμε. Πρέπει να σας πω ότι για να έχουμε αυτό τον ε, κύκλο, αν θέλετε, αυτή την, ε, τον ε, καλό κύκλο της οικονομίας, πρέπει να εφαρμόσουμε και πολιτικές σοβαρές εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω μία πτυχή συγκεκριμένα που αφορά τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Υπάρχουν πολλές πτυχές, κατά την άποψή μου, που έχουν αντιμετωπιστεί νομοθετικά, όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των πρώτων υλών που γίνονται όλο ένα και πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις δευτερογενείς πρώτες Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υπολογίσει ότι τα, τα 37 από τα 40 από 40 πρώτε ύλε, οι 37 έχουν, μειώσει τις, έχουν μειωθεί στι τιμέ. Αυτό ε, επηρεάζει και κυρίως ε, την ανακύκλωση των, ε, ηλεκτρον, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο πώς, τι θέλει να κάνει η Κομισιό όσον αφορά την ε, μείωση των, ε, της τιμής των πρώτων υλών, διότι με τον τρόπο αυτό ε, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη της αγοράς των δευτερογενών πρώτων υλών. Υπάρχει, ήθελα να κάνω και άλλη μια ερώτηση, ο προκάτοχός μου, ο συνάδελφός μου με προκατάλαβε, αλλά τέλος πάντων ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. που αναφέρει Φέρθηκε στην Καμόρα, στην, στην Καμπανία όμως ε, το πρόβλημα ε, δεν είναι οι αποτεφρωτές και η αποτέφρωση. Η, η Καμόρα δεν τα έκαιγε τόπου, ήθελε να τα εξάγει για να κερδίσει περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, ε, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε ε, ε, αυτά, τα, αυτές, ε, αυτά τα στερεότυπα και τις κοινοτυπίες που δεν ευνοούν κανέναν. Κυρία Κιώστιγκε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. με κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ και διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Εμείς τι βλέπουμε. Όλο και περισσότερο κονδύλια ευρωπαϊκά χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένα έργα που, αν τα δούμε εκ των υστέρων, στρέφονται κατά το δικό μας ε, καινοτόμων προθέσεων, πόσο μάλλον της κυκλικής οικονομίας. Αντιστρατεύονται δηλαδή τα δικά μας ε, έργα, τους στόχους και ακούμε και πολύ μεγάλη κριτική για τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς βλέπετε δυνατότητες χρηματοδότησης που να εγκρίνεται μόνο εφόσον συνάδων με τους στόχους και τους υλοποιούν τους στόχους αυτούς της κυκλικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία που πάνε σε τίποτα χωματερές. Τελείως λάθος κατεύθυνση. Και αυτό θα πρέπει να το βλέπουμε πάντα ως ενιαίο σύλλον. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να μην αφήνετε να σας προβοκάρει κανείς, από εδώ διάφοροι συνάδελφοι, που ζητούν το λόγο και θέλουν να κάνουν εντύπωση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για να είναι ο, ο, κόσμος σε καλύτερη κατάσταση αυτός που θα αφήσουμε. Και για τη σπατάλη των τροφίμων και τα απόβλητα από τρόφιμα, καλωσορίζω αυτό που λέτε, κάτι καλό σίγουρα θα βγάλουμε. Απλώς θέλω να πω ότι στα διαφορά κράτη-μέλη έχουμε πολύ διαφορετικές πραγματικότητες και ε, ε, μοντέλα υπολογισμού. Δηλαδή τα μετράνε με διαφορετικό τρόπο και τα ελοποιούν με διαφορετικό τρόπο τα προγράμματα για την αποφυγη αποφυγή σπατάλης τροφίμων. Γιατί φοβούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν φιλοδοξίες αλλά ε, παρεμποδίζονται να δρουν όσο θα ήθελαν. Καλά, υποστήριξη από διάφορες πλευρές εδώ που φωνασκούν δεν περιμένω, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει μόνοι μας να χειριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας και για την προθυμία σας να έρθετε εδώ και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Πίτρο που είναι εδώ μαζί μας. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τρεις καλές ειδήσει. Τον περασμένο μήνα ε, στο Βανκούβερ, ε, στον Καναδά, Είχαμε 24 ε, ορόφους ε, σε ένα ξύλινο ε, κτίριο και στη Βιέννη και στο Λονδίνο. Στο Χάκνη, στο Ανατολικό Λονδίνο, οικοδομήθηκαν λοιπόν τρία τέτοια ξύλινα κτίρια και αυτό είναι πολύ καλό γιατί έτσι περιορίζονται οι εκπομπές εξιδίου του άνθρακα και είναι πολύ καλό υποκατάστατο το ξύλο του ατσαλιού. Ε, του Χάλιβα. Επομένω, είναι καλό που υποκαθιστούμε ε, το, τον άνθρακα και τον Χάλιβα με ξύλο, τον πετόν. Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μακρόπνοο, όμως ε, κάποιες δεκαετίες στη συνέχεια μπορεί να ανακυκλωθεί. Και οι ξύλινες κουζίνες μπορούν να ανακυκλωθούν τέσσερις φορές και μετά το καλύτερο είναι βέβαια η αποτέφρωσή τους. Αυτό είναι πράσινη ενέργεια. Επομένω σα καλώ να λάβετε υπόψη την τεράστια ε, συμβολή που μπορεί να έχει το ξύλο στην ε, ε, βιώσιμη αυτή οικονομία και την κυκλική οικονομία που προτείνεται για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πολύ γρήγορα ένα ερώτημα για, τα, για τον κανονισμό για τα λοιπάσματα που εντάσσεται ε, στον σχεδιασμό για την κύκλική οικονομία. Αυτό που ζητούμε περισσότερο είναι βέβαια η εισαγωγή ορίων σχετικά με τις ε, ρηπαντικές ηρωπογόνες ουσίες. Αυτό θα εξάλληπτε ουσιαστικά τα περισσότερα από τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και παρά τα ξεκάθαρα ε, επιστημονικά στοιχεία ε, οδηγούμαστε σε αυτές τις λύσεις. Ποια είναι όμως η εναλλακτική. Πρώτον, ε, όμως θα είχαμε έτσι υψηλότερες εισαγωγέ από τη Ρωσία και τη Φιλανδία. Για τη Ρωσία τα πράγματα είναι αρκετά βέβαια γιατί ξέρουμε ότι ότι ε, η πλεονάζουσα εξόριξη θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις. Δεύτερον, νέες τεχνολογίες που να απομακρύνουν αυτές τις ε, ρηπογόνες ουσίες. Όμως αυτές είναι μόνο σε πειραματικό στάδιο. Είναι δύσκολο λοιπόν να βασιστούμε σε αυτές τις τεχνολογίες και δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις τεράστιες ποσότητες καδμίου ε, αν θα θέλαμε να το απομακρύνουμε. Και τρίτον, βιολογικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Πολωνία, ε, εντατικής γεωργίας δηλαδή. Όμως αυτό δεν ισχύει σε όλες ε, τις χώρες και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ε, περιορίζει τις εκπομπές αμμονίας και άλλων ουσιών δεν διευκολύνει την γεωργία. Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, λοιπόν, είστε βέβαιος ότι μπορείτε να διασφαλίσετε ε, την ε, επαρκή ποσότητα και παροχή λιπασμάτων σε μια καλή προσιτή τιμή στην αγορά ή μήπως θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ε, στρέβλωσης της αγοράς με το να στηρίζουμε συγκεκριμένους παρόχους και εποδιαστές σε αντίθεση με άλλους. Οι δικαιούχοι ουσιαστικά θα είναι αυτοί που θα προέρχονται από τη χώρα σας. Και κατά τη γνώμη μου, Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Βίτεμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θα ήθελα να ε, θέσω ένα ερώτημα για τον ε, κανονισμό και τα λοιπάσματα. Είμαι εισηγητή ε, στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων για αυτό το φάκελο. Συμφωνώ πλήρω με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλική οικονομία, για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση υλικών και ουσιών όπω το άζωτο και το καθεξής ε, και του φωσφόρου. Πρέπει να ανακτήσουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του φωσφόρου που χρησιμοποιούμε στη Γεωργία. Όμω, αν δούμε σε μεγαλύτερο βάθο το φάκελο, υπάρχει μεγάλη διασύνδεση με άλλε νομοθετικέ ε, διατάξει. Και φοβάμαι ότι οι στόχοι και οι προθέσεις είναι πολύ καλές όμως αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά σε ό,τι αφορά την επαξιοποίηση των βιολογικών, για παράδειγμα, λοιπασμάτων, εξαιτία άλλων νομοθεσιών. Γιατί δεν είναι βέβαιο ποιε θα είναι ακριβώς οι επιπτώσεις των άλλων νομοθετικών πλαισίων για την ε, ε, οδηγία για τα λοιπάσματα και ελπίζουμε να μην έτσι ε, αποτρέψουμε την χρήση των βιολογικών λοιπασμάτων. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια ή ε, να συνεργαστεί Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ αυτό για να υπάρξει μεγαλύτερη ε, σαφήνεια ω προ το αποτέλεσμα και για να δούμε ότι μπορούμε όντω να ανακτήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι ουσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πιετικάινεν. Mm. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν ε, θεωρώ ότι είναι ε, υπεύθυνο και δεν, δεν οφείλει να λογοδοτήσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, έναντι του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα κάνει ή δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για τα σχόλιά του για την ε, διεύρυνση του εφαρμογή ε, του οικολογικού σχεδιασμού στο μέλλον και εναρμόνιση των προποθέσεων για την επαναξιμοποίηση, την δυνατότητα ε, διόρθωσης επισκευής, ανακύκλωση και το καθεξής. Ε, ελπίζουμε αυτά να γίνουν όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και θετικά στοιχεία. Το δεύτερο που θα ήθελα ε, να αναφέρω και για το οποίο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω είναι η ενέργειά σας για το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ελπίζω πραγματικά ε, να υπάρξει βελτίωση του κανονισμού στο μέλλον, ούτω ώστε τα κονδύλια να διοχετεύονται μόνο σε τέτοιε επενδύσει που θα ε, τονώνουν την οικονομία. Άλλο στοιχείο τώρα για ε, τις δημόσιες προμήθειες, 20% του ΑΕΠ μας. Στην έκθεση του Κοινοβουλίου εκφράσαμε την επιθυμία μας να υποχρεωτικά να λαμβάνουμε υπόψη ε, την επαναξιμοποίηση των ε, υλικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε προταθεί στο Κοινοβούλιο και κατά την ε, εξέταση της σχετικής οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες. Είναι δύσκολο βέβαια να θεσπίσουμε τέτοιου είδους υποχρεώσεις και ελπίζω η αναθεώρηση της οδηγίας να καταστεί δυνατή κάποια στιγμή. Στο προσεχές μέλλον τουλάχιστον θα ήθελα να μας πείτε ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον ε, κλάδο αυτών των δημοσίων προμηθειών. Να γίνουν όλα αυτά δηλαδή υποχρεωτικά και να υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα. Ένα από τα εμπόδια που εντοπίζω εγώ είναι ότι δεν υπάρχουν γνώσεις, δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί για τις δημόσιες προμήθειες. Αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να πω. Αυτό είναι το επίγον ζήτημα σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα δικτών. Αν δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο δίκτυο δικτών, είναι δύσκολο να, να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το τομέα για να έχουμε εναρμονισμένους δικτές κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο χρόνος πιέζει και ένα βασικό θέμα που με απασχολεί είναι η διασπάθηση των τροφίμων. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λύση δεν υπάρχουν δείκτες, δεν υπάρχει κοινή μέθοδος σήμερα ε, που μπορεί να διευκρινίσει ε, αυτή την διασπάθηση των τροφίμων. Θέλω να ξέρω πού βρίσκεστε ε, αυτή τη στιγμή, τι, σε τι έχει καταλήξει η ομάδα εργασίες, που έχει σαν στόχο να μέχρι το 2030 να περιορίσει κατά 50% την σπατάλη των τροφίμων και ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της, υπερκατανα... της ε, διασπάθησης ε, βρίσκεται στο επίπεδο της κατανάλωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια εργαλεία έτσι, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για την ημερομηνία λήξης, για την ημερομηνία κατανάλωσης και μια και μιλάμε και για καταναλωτές κύριε Επίτροπε θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε αυτή την ε, παρέκκληση ε, τους ε, υφίστανται τα φρούτα και τα λαχανικά για να κρατήσουν περισσότερο μέσα στα ψυγεία. Αυτό δεν είναι ε, καλύτερη διαχείριση των ε, φρούτων και των λαχανικών, αλλά απλώς ένας, ένας άλλος τρόπος για να αυξήσουμε τα απόβλητα. Επίσης, θα ήθελα να δούμε τι θα κάνετε, πώς θα συνδυάσετε τα παλιά και τα νέα μέτρα όσον αφορά την περιβαλλοντική ετικετοθεσία, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν eco-labels αυτή τη στιγμή, γι' αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας, να μην δημιουργήσετε νέα μέτρα ή τουλάχιστον τα νέα μέτρα να είναι σε συμφωνία με τα υπάρχοντα, γιατί ε, η καλύτερη απλούσταυση, κύριε κυρία Αντιπρόεδρε, είναι ο σεβασμός των ήδη υφισταμένων μέτρων και η ίδια αντιμετώπιση. Η κυρία Κάινενμπακ. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση που είναι ίσως λίγο περιφερειακή σε σχέση με αυτά που σας απασχολούν. Αλλά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ε, θα πρέπει να συζητήσει το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας το αναφέρω. Και πρόκειται για τη συνέχιση της οδηγίας ε, FFH. Είναι μια οδηγία πάρα πολύ καλή ε, ως προς την νομοθεσία. για τους οικοτόπους αλλά το πρόβλημα είναι η υλοποίηση. Το είπαν και άλλοι και ο συνάδελφο ε, Φλόρενς και η κυρία Κιώστηγκερ μίλησε για χωματερές σήμερα. Ε, ανησυχούμε γιατί υπάρχει θέμα βιοπικιλότητας ε, και πολύτιμοι τόποι, είτε είναι υγρότοποι, είτε είναι λιβάδια, επειδή δεν θα χαρακτηριστούν ως πολύτιμοι για τη φύση, να χρησιμοποιηθούν, κινδυνεύουν ως χωματερές. Και στα πλαίσια του Refit δεν θέλουμε εμείς ε, να βαρύνουμε την οδηγία, ούτε να την ξανανοίξουμε, ούτε τίποτα. Απλώς να ενισχυθεί η εφαρμογή και η έλεγχη αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάμπους. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ που ήρθατε και μας ενημερώσατε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα έργα που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση των υδάτων, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους, έτσι λίγο πιο εκτενώς, γιατί τα αναφέρατε πολύ επιγραμματικά για το 2017. Επόμενη ερώτηση, πιο γενική, λαμβάνοντα υπόψη ότι είστε και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια, τι έχω δει. Κυκλική οικονομία, πράσινη οικονομία και σχέδια που έχουν οι δήμοι, κοινότητε, οι υπαρχίε, οι νομοί και οι αυτόνομε περιφέρειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ασχολείται με αυτό το θέμα, όχι μόνο νομοθετικά, αλλά και επικοινωνιακά. Μιλήσετε για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το έψι, δηλαδή, υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενισχύσεις, αλλά δεν ξέρουν τι έχουν πάρει και από πού. Ε, και επειδή υπάρχει κρίση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν δίνει αποτελέσματα, ε, πέρα από την νομοθετική δουλειά που είναι δικιά μας βεβαίως, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω, να κάνει κτήμα της και αυτή τη συζήτηση και στο επικοινωνιακό, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στην κυκλική οικονομία. Είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα τελευταίο. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό να περάσει έτσι. Η δουλειά μας δεν είναι να επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να προωθούμε για να υπάρχει συνεργασία η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επικοδομητική και είναι και καλόπιστη. Και αν είναι κακόπιστη δεν αξίζει καν να ασχοληθείτε, ούτε να πικραθείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Ο κύριος Νταντά σε ένα από τα θέματα τα οποία μας αφορούν, μας απασχολούν στην κυκλική οικονομία υπάρχει ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό που είναι το νερό. Το νερό εμπλέκεται στην δραστηριο, ανθρώπινη δραστηριότητα, στη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Όμως η αρχή της κυκλικής οικονομίας ε, έχει σαν στόχο να επαναχρησιμοποιήσει, να ανακυκλώσει ε, τα προϊόντα. Αυτό χρησιμοποιείται πολλές φορές για το νερό, όμως δεν μιλάμε για τη χρήση του νερού σαν απόβλητο. Το Κοινοβούλιο όμως έχει ζητήσει σε μια πρόσφατη έκθεση ε, να υπάρξει μια νέα νομοθεσία για τα, για νερά, για τα λίματα. Όμως ε, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα και έχουμε, θέλουμε μία πρόταση λεπτομερή για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα λίματα για πότισμα, για ε, άρδευση κτλ. Βέβαια, θα πρέπει και στην βιομηχανική διαδικασία να μειώσουμε την κατανάλωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε μέσω του προπολογισμού για την ε, έρευνα να δώσει κάποια κίνητρα στην βιομηχανία, στην οικονομία γενικότερα, να υιοθετήσει διαδικασίες ε, που να εξοικονομούν νερό. Το περιβαλλον... η... η αλλαγή του κλίματος δεν αφορά μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά αφορά και την Ευρώπη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα απευθυνόμενη στον Αντιπρόεδρο Κατάιναν να μιλήσω και θετικά σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία. Στην Ολλανδία το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης, είναι το πρόβλημα η πολιτική. Οι υπουργοί είναι αυτοί που κάνουν τους ανήξερους, ενώ η οικονομία, ο κλάδος είναι αυτός που ε, το έχει σηκώσει τα μανίκια. Και νομίζω ότι ε, μάλιστα θα υπάρξει μια συνδιάσκεψη του χρόνου στη χώρα μου, ακριβώς και αυτό το σημείο, συγγνώμη. Όπως αναφέρατε κι εσείς λοιπόν, ε, δεν είναι μόνο δικό του θέμα, είναι δικό μας των πολιτικών δηλαδή. Ε, συμφωνώ εδώ με τον κύριο Χάτεμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο σε ό,τι αφορά ε, τα ορυκτά και αυτές τις ουσίες ακούω από επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν ότι πρέπει να επενδύσουν 100 εκατομμύρια για να λάβουν ε, ε, κονδύλια από το ΕΦΣΥ. Δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί άλλα έχουμε ακούσει από εσά. Ε, και μιλούμε για την αξιοποίηση του φωσφόρου. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να εργαστούμε επί μιας ε, πλατφόρμας επενδύσεων σε ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίηση ορυκτών. Στην Ολλανδία το 1 τέταρτο των αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει να κλείσουν μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας ε, των ε, αζωτούχων. Εγώ είμαι υπέρ των περιβαλλοντικών νομοθεσιών, όμως Όπω είπε και ο Επίτροπο ε, Χόγκεν, είπε ότι θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε θετικέ διατάξει. Ακούσαμε αρνητικέ ε, κριτικέ για την Ολλανδία. Εμεί ε, συνεχίζουμε την προσπάθειά μα. Ε, νομίζω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά και στο μέλλον πιο συγκεκριμένα να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τα ερωτήματά σας. Το λόγο έχει ο κύριος Αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές ερωτήσεις και πολύ άρθμες. Η κυρία Γκροστέτ έθιξε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να απαντήσω. Έχω ακούσει και εγώ ακριβώς την ίδια είδηση ότι τα πλέον ε, μοντέρνα και συγχρονισμένα ευρωπαϊκά ελαστικά που κατασκευάζονται από ε, σύγχρονα υλικά είναι κάποιες φορές πιο ακριβά σε σχέση με τα κινέζικα κτλ. που κατασκευάζονται από παρθένες πρωτεσίλες. Όμως δεν ξέρω τι να, κάνω, τι να κάνουμε, εκτός από το να βελτιώσουμε ε, τον ανταγωνισμό και να μειώσουμε τις τιμές. Δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στην ίδια γαλλική επιχείρηση που τα κατασκευάζει. Έχω ακούσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου η εταιρεία με leasing παρέχει τα ελαστικά στα αεροσκάφη. Επομένω, ε, απλώς με leasing ε, εφοδιάζει ε, τις απογειώσεις και προσγειώσεις, το οποίο λειτουργεί καλά ως μοντέλο και έτσι μπορούν να, τις, να επαναχρησιμοποιήσουν τα ελαστικά γιατί ε, είτε τα χρησιμοποιούν εκ νέου είτε τα μεταπολούν σε άλλου πελάτε του. Το leasing λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια συγγνώμη, βράχη πρόθεσμη λύση σε κάποιου ε, τομείς, όχι όμω στον τομέα στον οποίο αναφερθήκατε εσεί ίσω. Καλύτερη αγορά λοιπόν και αύξηση της ζήτησης από τους καταναλωτές. Ίσως αυτό να ήταν η πιο βιώσιμη λύση. Επίσης θα μπορούσαμε να θέσουμε ε, πρότυπα σε ό,τι αφορά την ε, κατασκευή ελαστικών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ίσο πεδίο ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές. Αυτό θα ήταν μια άλλη λύση. Μια παρόμοια ερώτηση αφορούσε το κόστος των παρθένων πρώτων που είναι πολύ χαμηλές. Ιδίω οι τιμέ του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλή ε, και έτσι αυτό παρεμποδίζει ε, τι επενδύσει. Και δυσχεραίνει τη χρήση των ε, δευτερογενών πρωτονυλών, όπω το πλαστικό. η καλύτερη αλλά πλέον δύσκολη λύση είναι να ε, κοστολογούμε πιο αποτελεσματικά τον, ε, τις εκπομπές άνθρακα από ό,τι κάνουμε σήμερα. Η τιμολόγηση αυτή θα ήταν η λύση για όλα μας τα προβλήματα ουσιαστικά, ιδίως ε, για τις περιβολητικές προκλήσεις. Γι' αυτό η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ε, τιμολόγηση του, των εκπομπών άνθρακα. Οποιαδήποτε άλλη λύση που βασίζεται στις επιδοτήσεις δεν είναι βιώσιμη. Είναι λοιπόν απαραίτητε οι προσπάθειε ε, αύξηση τη τιμή των εκπομπών του άνθρακα. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα των πλαστικών. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία εντός των υπηρεσιών μας, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούν λοιπόν οι υπηρεσίες μας να δουν πώς ε, μπορούμε ε, να προετοιμάσουμε, να προλιάνουμε το έδαφος για τη στρατηγική για τα πλαστικά. Ο δικός χάρτης που προκύπτει από, αυτό, από αυτή την υπηρεσιακή διαδικασία θα είναι σύντομα διαθέσιμος και ελπίζουμε μέχρι τον Ιανουάριο να έχει δημοσιοποιηθεί. Τότε λοιπόν θα γνωρίζουμε ε, ποια είναι τα πρώτα βήματα ε, τα οποία θα κάνουμε για να προετοιμάσουμε τη στατική για το πλαστικό. Αν δείτε λοιπόν τη στρατηγική ε, περιαποβλήτων, είναι εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα και υπάρχουν πολλές θετικές γωνίες. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική για τα πλαστικά. Όλοι συμφωνούν για τους ε, στόχους, αλλά όταν περνάμε στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων ε, και την διερεύνηση διόδων, τα πράγματα δυσκολεύουν δεν υπάρχει καμία υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να θέλει να μπλοκάρει, να παρεμποδίσει την ε, ε, κατάρτιση αυτής της ε, στρατηγικής για το πλαστικό, απλώς χρειάζεται χρόνος. Τώρα, για τις σπατάλη τροφίμων. Υπήρξαν αρκετά σχόλια και ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Σίγουρα γνωρίζετε καλά την πρόταση με την υποχρέωση ανάληψης ενεργειών και πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της πατάλης τροφίμων. Ε, η εισηγήτρια κυρία Μποναφέ πρότεινε να συμπεριλάβουμε έναν ορισμό της σπατάλης τροφίμων και σχετικών στόχων μείωσης της σπατάλης. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας ε, ρώτησαν ακριβώς ε, τι συμβαίνει με αυτούς ε, τους στόχους. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει ε, μία βασική γραμμή ούτε ένας μηχανισμός παρακολούθησης. Είναι εύκολο να θέσουμε έναν... Ε, θα ήταν εύκολο να θέσουμε έναν στόχο αν γνωρίζαμε από πού προκύπτει αυτή η σπατάλη τροφίμων, ποια είναι αυτή η βασική γραμμή, η baseline και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο μηχανισμό παρακολούθηση. Γι' αυτό και ένα ε, νομικά δεσμευτικό στόχο είναι δύσκολο να οριστεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να γίνει αυτό στο μέλλον. Στο σχέδιο δράσης μας αναφέρεται ότι φέτος πρέπει ε, να αναλάβουμε κάποιες ενέργειες για αυτό το τομέα. Πρώτον, θέσπιση μιας νέας πλατφόρμας όπου κράτη-μέλη και άλλοι ε, φορείς ε, στην επιστική αλυσίδα ε, θα συνεργάζονται για να βρουν τρόπους επίτευξης του στόχου για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το καθεξής. Έχει δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα την 1η Αυγούστου και θα τεθεί σε λειτουργία πολύ σύντομα θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα αυτή η πλατφόρμα για τον εντοπισμό προβλημάτων και την εξέβρεση λύσεων. Στο φετινό πρόγραμμα εργασιών επεξεργαστήκαμε και μια κοινή ορολογία για την μέτρηση του επιστημισμού, συγγνώμη, της πατάλης τροφίμων. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και να μας βοηθήσει να θέσουμε στόχους και το πρώτο προσχέδιο θα τα εξετάσουμε στην πρώτη συνάντηση της πλατφόρμας το Νοέμβριο. Θέλουμε να διευκρινίσουμε και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε σχέση με τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, να διευκολύνουμε την, ε, τη δωρεά τροφίμων. Σε αυτά τα ζητήματα θα έχουμε και ευρωπαϊκές κατευθύνες γραμμές και το πρώτο προσχέδιο θα το εξετάσουμε στην πρώτη συνάντηση της πλατφόρμας. Η τελική υιοθέτηση θα γίνει στα τέλη της επόμενης χρονιάς. Κατευθύνες γραμμές τώρα για, την, για να διευκρινίσουμε το νομικό καθεστώς ε, των ε, τροφίμων που ε, οδηγούνται προ τι ζωοτροφέ. Έχουμε διαβουλεύσεις μεταξύ τη Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων και της Διτσισάνκο και θα ολοκληρωθεί του χρόνου αυτή η διαδικασία. Επομένω, υπάρχουν διαδικασίε ε, εντό των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλώ ε, παίρνουν χρόνο. Βεβαίω, θα πρέπει να καταλήξουμε σε, από τα αποτελέσματα. Τώρα, μια συνεκτική προσέγγιση σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για την αποτέφρωση και το καθεξής, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να βρούμε πολλές, να εξετάσουμε μάλλον πολλές οδηγίες, πολλές προτάσεις, ε, στόχοι για την κυκλική οικονομία, για την χρήση γης, για την ε, βιοοικονομία, ενεργειακή απόδοση όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε συνεκτικά. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά συμφέροντα που παίζουν εδώ και πολλά διαφορετικά τέτοια συμφέροντα. Επομένω, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής, είναι τεράστιο οικονομικό ζήτημα. Εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, απόψεων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δημιουργεί τεράστιες πιέσεις για εμάς. Πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε μακρόπνο σχεδιασμό ε, και να θεσπίσουμε εύλογα πρότυπα και κανονισμούς. Ξύλινα κτίρια, σας ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ξύλινη καμπίνα σε ένα δάσο και πάντα μου αρέσουν αυτά τα ξύλινα κτίρια. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. μου δημιουργεί έκπληξη που δεν αξιοποιείται περισσότερο το ξύλο στην Ευρώπη στα κτίρια. Νομίζω ότι ε, στην Ιαπωνία αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο και εισάγουν μάλιστα ευρωπαϊκή ξυλία για ε, την οικοδομή τους, τις κατασκευέ τους. Θα πρέπει και εμείς ε, να κάνουμε το ίδιο. Κανονισμός λοιπασμάτων. Πολύ καλά τα σχόλιά σας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε ζητήματα υγείας. Εδώ το πρόβλημα είναι το κάδμιο και άλλες ε, τοξικές, τοξική ρήπη. Δεύτερον, δύο κύρια ζητήματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του κανονισμού λοιπασμάτων. Πρώτον, να περιορίσουμε τα επίπεδα καδμίου για λόγους ε, δημόσιας υγείας. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα νέο ε, περιβάλλον αγοράς για τα βιολογικά λοιπάσματα. Κατανότα όσα λέτε. Αν υπάρχουν άλλοι κανονισμοί που αποτρέπουν τη χρήση βιολογικών ε, ουσιών κατά την ε, παραγωγή λιπασμάτων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ένα, μια από αυτές τις καινοτόμες ε, συμφωνίες που αναφέρατε. Πρέπει λοιπόν να το ε, εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, πώς θα δημιουργήσουμε μία αγορά για τα βιολογικά λοιπάσματα. Οι φωσφορικές ε, ενώσεις. Ξέρετε ότι είναι σπάνια πρώτη δεν θα αντέξει για πάντα και ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για μας για να βρούμε νέους τρόπους μέσω της ε, οδηγίας. Πράγματι, η Ρωσία και η Φιλανδία μπορούν ε, να παραγάγουν καλύτερες ε, τέτοιες ενώσεις στο μέλλον, προς το παρόν μάλλον, αλλά αυτό δεν είναι μια βιώσιμη λύση για το μέλλον. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπάσματα και για να δοθεί πρόσβαση μάλλον στο μέλλον στην αγορά θα πρέπει να συμμορφούνται κανείς με τα χαμηλότερα επίπεδα καδμίου. Αν θέλει να χρησιμοποιεί κανείς λιπάσματα που δεν συμμορφούνται με τα επίπεδα καδμίου να τα ε, παράξει λοιπόν στην αγορά του αλλά δεν θα έχει πρόσβαση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά λοιπόν για να έχουμε μια καλύτερη ενιαία αγορά για τα βιολογικά λιπάσματα η πρότασή μας νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους προβληματισμούς που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αυξήσει την τιμή των λοιπασμάτων. Τουλάχιστον όχι μεσοπρόθεσμα. Γιατί όσο περισσότερα λοιπάσματα υπάρχουν στην αγορά, τόσο θα πέσει η τιμή. Δημόσιες προμήθειες. να διαβάσω μια στιγμή τι είπατε. Έχουμε νέες κατευθύνες γραμμές, όπως ξέρετε, για αυτό το ζήτημα. Δεν είναι υποχρεωτικά αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή, όμως ε, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνική αρρωγή στα κράτη-μέλη για να αξιοποιούν τις νέες κατευθυντήρες γραμμές για τις πιο πράσινες δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να λαμβάνει κανείς υπόψη τη δυνατότητα χρήσης ανανεώσιμων υλών ή υλών που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίησή του στις δημόσιες προμήθειες. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ίσως στο μέλλον να είμαι σε θέση να προσθέσουμε κάτι στι κατευθυντήριε γραμμές. Ο οικολογικό σχεδιασμό, συγγνώμη, η οικολογική επισήμανση ε, είναι στη διαδικασία ρήφητα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί ή όχι. Όμως, ε, συμφωνώ με τις επιφυλάξεις ότι όταν θα έχουμε πολλά οικολογικά σήματα στην αγορά ε, θα δημιουργηθεί σύγχυση στους καταναλωτές και δεν θα πιστεύονται κανένα. Επομένω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό τον τομέα γιατί ε, τα, τα, οικολογικά σήματα που έχουν αυτή τη στιγμή γίνονται ευρέως αποδεκτά και από τους καταναλωτές και από τον κλάδο και από τις ενώσεις καταναλωτών. Επομένως, δημιουργείται και εμπιστοσύνη στην αγορά. πλατφόρμες για την ε, χρήση των ε, ορυκτών και αυτό θα ήταν μια καλή λύση για την ανταλλαγή απόψεων και τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, ίσως και για να βρούμε νέους ε, τρόπους να επενδύσουμε σε αυτόν τον κλάδο. Υπήρχε ένα ακόμα ερώτημα για το ΕΦΣΥ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει αυτό που αναφέρεται με κάποια κράτη-μέλη που τα κατά τη κυκλική οικονομία. Εγώ προσωπικά δεν ε, έχω δει μεγάλα ε, τέτοια προγράμματα διαχείρισης ε, αποβλήτων που να προσπαθούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ. Ίσως να είναι τόσο επικερδή αυτά τα προγράμματα που να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την αγορά, αλλά δεν νομίζω. Επομένω, θα πρέπει να διαβιβάσουμε και το μήνυμα στα κρατημέλη μας ότι υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο που μπορεί να χρηματοδοτήσει ε, νέες τεχνολογίε που είναι πιο ε, σε σχέση με παλαιότερε. και έτσι να αντικαθιστούν άλλα παλαιότερα τέτοια προγράμματα. Κλείνοντα ένα τελευταίο σχόλιο ε, για την οδηγία που βρίσκεται υπό fitness check, Nature Directive. Υπάρχει τεράστια πίεση από τη δημόσια, την κοινή γνώμη να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτού του fitness check. Δεν έχω δυστυχώς κάτι να προσθέσω εδώ συνεχίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε τα αποτελέσματα από το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much to you for your... Εγώ σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Μπορούμε τώρα να τελειώσουμε με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και να περιμένουμε ένα λεπτό για να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο 16. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Γκουίντο Ράζη, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, εν ώψη του τακτικού διαλόγου που έχουμε με τον ΕΟΦ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσουμε και διοργανώνουμε κάθε χρόνο μια επίσκεψη του εκτελεστικού διευθυντού, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συζητούμε και ε, ε, το πρόγραμμα της εργασίας το 2016 και πώς αυτό εντάσσεται στο πολιετές μέχρι το 2020. Όσοι ήθιστε θα ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση του κυρίου Ράζη και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο ε, στο σύνδεσμό μας την κυρία Μπούρζαν και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κύριε Ράζη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να μπω κατευθείαν στο ψητό, <laughs> στο ταμπού μάλλον, που είναι το Brexit και οι πιθανές συνέπειες του στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Έχουμε έναν άμεσο αντίκτυπο και αυτό είναι το κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας που ζούμε ήδη. Το άλλο θέμα είναι ενδεχόμενη επαγκατάσταση του ΕΟΦ κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχούμε βαθύτατα ότι έτσι θα χάσουμε πολλούς ε, εμπειρογνώμονες και προσωπικό, πολύτιμο. Και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και να προκαλέσει προβλήματα, ε, γιατί έχουμε 4.000 εμπειρογνώμονες που συνδέονται ε, στο δίκτυό μας ε, και γενικότερα ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να εξακολουθούμε να δίνουμε την ε, ποιότητα που παρέχουμε σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. 98% ναι, είναι η συμμόρφωσή μας και αυτό το επίτευγμα έρχεται σε ένα πολύ περίπλοκο σύστημα. 36.000 επισκέψεις έχουμε ε, εμπειρογνωμόνων και συνέδρων που θα πρέπει να έρχονται το σωστό χρόνο με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα σε πολύ συγκεκριμένες ώρες κτλ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκος ο μηχανισμός που είναι σαν γραμμή παραγωγής εργοστασίου ουσιαστικά. position ε, και ανησυχούμε γιατί θα πρέπει να είμαστε και στο ανάλογο περιβάλλον όπου να υπάρχει και η διασύνδεση αυτή that we και μια πολυπλοκότητα που πρέπει να διαχειριστούμε. Αλλά ας πάμε σε κάποια πιο θετικά και πολύ θετικά. Στις 20 Οκτωβρίου για πρώτη φορά ε, στη νέα μας ιστοσελίδα δημοσιεύσαμε τα ε, στοιχεία κλινικών δοκιμών για δύο νέα φάρμακα τα οποία εγκρίναμε ήταν πολύ μακρύ το ταξίδι, τεσσάρων ετών και με την σταθερή και μόνιμη υποστήριξη της δικής σας Επιτροπής ε, καταφέραμε. Και περιμένουμε ε, πολλά θετικά και ευεργετήματα σε πολλά επίπεδα θα είναι προς όφελος και των ερευνητών και των εργαζομένων ε, στον χώρο της υγείας, ε, καθώς επίσης και θα έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη και από πλευρά των ασθενών προς τους θεσμούς. Ε, τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιταχύνουν την καινοτομία, να μειώσουν τις επικαλύψεις και τους κινδύνους. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την πρωτοβουλία αυτή που έχει διαμορφώσει μια παγκόσμια συζήτηση και τελικά ε, και ε, ο κλάδος η φαρμακοβιομηχανία έχει γίνει πολύ συνεργάσιμη. Οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να σας πω ότι να φοβούνται τώρα την ε, υπόθεση αυτή και το ρίσκο χαίρονται για τις δυνατότητες που παρέχονται. Ε, υπάρχει κάποια επίκριση ως προς τη διαφάνεια μας ε, και έχουμε δεχτεί και προσωπικές επιθέσεις και εμείς όλα αυτά απαντούμε με γεγονότα. Περίπου 250.000 σελίδες έχουμε δημοσιεύσει και μόνο δύο από αυτές ε, είναι για ε, λόγους εμπορικούς, ενώ 10.000 έγγραφα έχουν επίσης ε, κατεβαστεί από το διαδίκτυο τις τελευταίες τις εβδομάδες. Εσείς εγκρίνατε μια νομοθεσία το 2010 που μας έδωσε μεγάλο και πολύ ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των φαρμάκων. Άρχισε το 2012 η εφαρμογή και έτσι καταφέραμε να ε, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον αντίκτυπο των ουσιών αυτών και τώρα είμαστε σε καλύτερη μοίρα να ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα. Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Υπάρχει μια επιτροπή για φάρμακοεπαγρύπνηση που λέγεται PRAC και κάθε χρόνο περίπου 100 ε, σημεία ελέγχει και κάνει 600 εκτιμήσεις κινδύνου για ε, δραστικές ουσίες. Αυτά όλα εκ των προτέρων, έτσι προληπτικά, για να δούμε πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να διαχειριστούμε και τους γνωστούς και τους αγνώστους κινδύνους και το ρίσκο. Και έτσι να αντιδρούμε καλύτερα. Επιπλέον, ε, αναφέρονται οι παρενέργειες από τους ίδιους τους ασθενείς σε ποσοστό που αυξήθηκε πάνω από 50% και η Επιτροπή ε, ε, παρέπεμψε 31 περιπτώσεις ασφάλειας και έτσι ε, ώστε όλοι οι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την ίδια προστασία. Τώρα λοιπόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση για να δρούμε γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, να προστατεύουμε το κοινό με κάποιους περιορισμούς ή ακόμα και αναστολή αδειών ή καλύτερη ε, καθοδήγηση για την καλύτερη χρήση του φαρμάκου. Η προστασία βεβαίως των ασθενών από τις επιβλαβείς συνέπειες και παρενέργειες είναι ένα στοιχείο της ε, δράσης μας και της ευθύνης μας. Ε, Βεβαίω χρειάζεται και επιγόντω να βρούμε νέε θεραπείε και νέα φάρμακα για ασθενεί που περιμένουν με πολλέ ασθένειε. Κατά τη διάρκεια του ενεστώτο έτου έχουμε ολοκληρώσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με διάφορους φορείς ε, εκτίμηση τεχνολογίας υγείας και έχουμε λανσάρει το, το Prime που είναι ένα νέο σχήμα ε, για την υποστήριξη νέων ε, φαρμάκων χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια και στις προδιαγραφές μας. Βεβαίως αυτό αφορά μόνο για φάρμακα που έχουν στόχο συγκεκριμένες έτρικες ανάγκες. Έτσι ε, έχουμε καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερο προγραμματισμό. Τι σημαίνει καλύτερος προγραμματισμός. Ε, μπορούν οι εταιρείες να παράγουν στοιχεία και δεδομένα υψηλή ποιότητα, καλύτερη πρόσβαση και πιο αξιόπιστα στοιχεία για την αξιολόγηση των φαρμάκων. Και καλύτερο σχεδιασμό σημαίνει χαμηλότερο ρίσκο ε, στους ασθενείς που υπόκεινται στι κλινικές μελέτες, τις υφίστανται δηλαδή, και ε, να μην υπάρχει έκθεση σε άχρηστε επιπλέον ε, κλινικές δοκιμές. Αυτό που θα ήθελα να σας αναφέρω τώρα, το τελευταίο πρόβλημα που έχουμε είναι η αηφορία και η βιωσιμότητα του δικτύου μας γιατί αλλάζει η κατάσταση, αυξάνεται ο φόρτος. παραδοσιακά η αξιολόγηση των φαρμάκων γίνεται από ε, μία ομάδα, από ένα κράτος μέλος. Παρόλο που ε, η νομοθεσία έχει στο μυαλό της ένα πολυεθνικό σχήμα. Τώρα υποστηρίζουμε πολυεθνικά τέτοια σχήματα, δηλαδή ε, υπάρχει ένα συντονιστή που είναι ένα κράτος μέλος, αλλά εκεί μπορεί να συνεργάζονται οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες, οι καλύτεροι ειδικοί από όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο από ένα κράτος. Αυτή η πολυεθνική λοιπόν ομάδα και αντίληψη ε, έχει επιτύχει πάρα πολύ. 24 κράτη-μέλη συμμετέχουν, είναι το πιο ψηλό επίπεδο που είχαμε ποτέ και βεβαίως ε, αυτό θα είναι πολύ πιο κρίσιμο καθώς ε, κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλούς εμπειρογνώμονες με το Brexit. Και βέβαια αυτό τι δείχνει, ότι η επιστήμη δουλεύει καλύτερα χωρίς σύνορα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή σας, πρώτα απ' όλα για την πάγια υποστήριξη ε, ε, για την έγκριση του προπολογισμού μας, αλλά όχι μόνο, και την υποστήριξη για επιπλέον χρηματοδότηση από το Συμβούλιο. Έχουμε πρόβλημα τεράστιο με τη μείωση των ανθρωπίνων πόρων, γιατί έχουμε περισσότερο έργο και πιο σφιχτά χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες και θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιδείτε η ποιότητά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα ήθελα επευκαιρία να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τον Γκρότε για την καλή συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν. Πάντα ήταν προσιλωμένο ε, στην προσπάθεια αυτή και στη βοήθεια προς εμάς. Και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι αναλαμβάνει τώρα η κυρία Μπιλιάνα Μπόρζαν ε, από τον κύριο Γκρότε και θα είναι ο σύνδεσμός σας με τον ΕΟΦ. Και σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω να συνεχίσουμε την καλή και αγαστή συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now we can... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση ακούγοντας πρώτα το σύνδεσμό μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ καθηγητή, κύριε Ράζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ για να μας ε, κάνετε μια παρουσιανική παρουσίαση των ε, επιτευμάτων της ΕΜΑ την τελευταία χρονιά. Θα ήθελα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Φαρμάκων. Ε, θα ήθελα να ε, πω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και ο προκάτοχός μου έκανε εξαιρετική δουλειά και πραγματικά νομίζω ότι θα συνεχίσω και εγώ την τόσο καλή συνεργασία γιατί ούτως ή άλλως ο Ευρωπαϊκός Ευρωπαϊκός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, θα περνάει δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προβλέπετε σαν πιθανές αρνητικές συνέπειες του Brexit στον ΕΟΦ, έστω και πριν από την επανεγκατάσταση, την μετακόμιση του ΕΟΦ. Υπάρχουν λειτουργικές δυσκολίες και αν ναι, πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Μια και κανείς πραγματικά δεν γνωρίζει πώς θα διεξαχθεί το Brexit. Ε, έχετε εργαστεί με βάση κάποια σενάρια. Μια και πολλοί σε αυτή την αίθουσα ενδιαφέρονται για το πώς θα γίνει η μετακόμιση του ΕΟΦ, μήπως θα μπορούσατε να μπείτε σε κάποιες λεπτομέρειε. Πότε θα πρέπει να μετακομίσει, πριν ή μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν ε, προβλήματα στην ε, λειτουργία του ΕΟΦ λόγω της μετακόμισης. Επίσης, ε, ήθελα να ρωτήσω εσείς έχετε λόγο για το ποια θα είναι η μελλοντική σας έδρα. Το Brexit ε, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα που έχει τεθεί μέχρι στιγμής. Βέβαια όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα και δεν είναι το μόνο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το 2015 ο ΕΟΦ έκανε μία έκθεση για τις ε, ε, συμφωνούσε, που αφορούσε δύο σύνδρομα, κυρίως σε νέες γυναίκες που είχαν κάνει το εμβόλιο για το... How often does EMA ε, contact referral of... Το HPV. Ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα εμβόλια έχετε κάνει έρευνες, θεωρήσατε ότι είναι ένα προϊόν που δεν είναι ασφαλές. Επίσης, ε, οι συνέπειες για τον αυτισμό. Έχει καμιά συνέπεια, υπάρχει κάποια παρενέργεια, αν θέλετε. Και επίσης, ε, ποιες, ε, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για την διαδικασία εμβολιασμών. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μέλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. δεν είδα τον κατάλογο εδώ. Η κυρία Γκροστέτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω στο διευθυντή, τον κύριο Γκουίντο Ράζη, ότι είναι μεγάλη ευχαρίστηση πραγματικά να τον συναντάμε κάθε φορά και να συζητάμε μαζί του και θα ήθελα μέσω αυτού να εκφράσω την υποστήριξη προς όλο τον οργανισμό, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά κατά από δύσκολες συνθήκες, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάμε όλο, ένα και περισσότερα πράγματα από τον ΕΟΦ, χωρίς να του χορηγούμε τα απαραίτητα μέσα. Δύο σημεία θα ήθελα να συζητήσουμε. Καταρχάς το ένα αφορά τη νέα διαδικασία έγκρισης των φαρμάκων. Αυτή η διαδικασία ε, στοχεύει σε θεραπευτικές, σε θεραπευτικά πεδία όπου μέχρι στιγμής η ιατρική αντιμετώπιση δεν είναι ικανοποιητική και στηρίζεται σε μία προωθημένη αν θέλετε διαδικασία και που στηρίζεται και σε φάρμακα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην ε, αγορά. Αυτό καινοτόμα φάρμακα και αυτό είναι καλό διότι οι ασθενείς έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα εφόσον ε, υπάρχει ανάγκη, όμως υπάρχουν και κάποιες σκιές, κυρίως όσον αφορά την ενημέρωση και την προστασία των ασθενών. Θα ήθελα να με καθισχάσετε λιγάκι αν γίνεται. Ο οργανισμός έχει δημοσιεύσει μια εξαιρετική έκθεση φέτος το καλοκαίρι για την αξιολόγηση του προγράμματος, του πιλωτικού αυτού προγράμματος και δεν ήθελα να ξέρω ποια είναι η συνέχεια που θα δώσετε σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Δεύτερο σημείο, δεύτερο σημείο το Brexit βέβαια, και εδώ θα ολοκληρώσω γρήγορα γιατί ούτως ή άλλως το αναφέρατε και εσείς και η συνάδελφός μου, το Brexit ε, όντως ε, είναι μια, ένα, μια πηγή ανησυχίας για όλους, μια ανησυχία, πηγή ανησυχίας για αυτούς που εργάζονται και θα ήθελα όντως να γίνει μια μετακόμιση κάτω από τις καλύτερες ε, δυνατέ συνθήκες προς όφελος του οργανισμού βέβαια και θα ήθελα να μου πείτε εσείς ε, πώς ε, βλέπετε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, θεωρείτε της μετακόμισης. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στον οργανισμό και με την ε, σύμφωνη γνώμη της ε, Λιόν, από την οποία προέρχομαι, ε, θα προτείνω η Μητρόπολη αυτή να υποδεχθεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, διότι ούτως ή άλλως είναι γνωστό το κλίμα που επικρατεί και το περιβάλλον το ιατρικό, αν θέλετε, της περιοχής. Ευχαριστώ κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς εσάς. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά τους υπερβολικούς ε, κανονισμούς ε, προσωπικών δεδομένων ε, για τις καινοτομίες που άπτονται των ευρυστεχνίων στα φάρμακα. Η σημερινή νομοθεσία επιτρέπει στις φαρμακοβιομηχανίες να πατεντάρουν νέα προϊόντα που ουσιαστικά είναι παλιά προϊόντα με ορισμένες τροποποιήσεις μόνο και μόνο για να επεκτείνουν ε, την ε, διάρκεια προστασίας των προϊόντων αυτών. Τα δικά μας στοιχεία μας δείχνουν ότι έως και 80% των νέων φαρμάκων εντός αγωγικών δεν είναι και τόσο καινούργια τελικά. Και όμως πάλι πατεντάρονται αυτά τα φάρμακα και πολλούνται υπό ε, το κοστολόγιο αυτό που αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν. Ποια είναι η δική σας γνώμη λοιπόν για τη σημερινή ισχύουσα νομοθεσία. Το δεύτερο ερώτημα αφορά κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας, την πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα. Είπατε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτή είναι η δική σας γνώμη. Από την άλλη, βλέπουμε ότι εξαιτία των ε, παράλληλων επανεξαγωγών βλέπουμε πλέον ότι σε πολλές χώρες από σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα γιατί αυτά τα φάρμακα μεταπολούνται αλλού. Γιατί θεωρούνται εμπόρευμα τα φάρμακα. Και έτσι τα κράτη-μέλη και οι εθνιστικοί φορείς δεν έχουν και άλλες ε, επιλογές. Ποιος Ποια είναι η γνώμη του ΕΟΦ. Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση. Υπάρχουν μέσα και τρόποι ε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο που δυστυχώς υπάρχει. Και αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Και αυτό δεν είναι θέμα ε, ελεύθερης αγοράς. Ευχαριστώ κυρία Αουκέν. Γεια σας κύριε Ράζη και καλωσορίσατε. ορίσατε. Χάρηκα που αναφερθήκατε στη διαφάνεια για στις κλινικές δοκιμές και ότι προσβλέπετε στο να ε, υπάρξουν ε, καλά αποτελέσματα μετά από αυτή τη μακρά διελκυστή με την ε, φαρμακοβιομηχανία. Έχω μερικά προβλήματα με τη διαφάνεια. Πρόσφατα ο ΕΟΦ ξεκίνησε μια διαδικασία για τη σύγκρουση συμφερόντων για να τα ελέγχετε. Πόσους πόρους έχετε και πόσους ανθρώπους ε, για τους εμπειρογνώμονες, πώς τους ελέγχετε για τη σύγκρουση συμφερόντων και έχετε εντοπίσει περιπτώσεις ανελικρινών δηλώσεων ε, σύγκρουση συμφερόντων και αν ναι, πώς το χειρίζεστε αυτό. Όταν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής ε, διαχείρισης και διοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν αρκεί κάποιος να δηλώνει ε, για μια σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ πρόκειται για σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή και την υγεία των πολιτών και των ασθενών. Ξέρετε ότι έχουμε κάπως απογοητευτεί από τη στρατηγική σας για την έρευνα. Ε, ε, αναφέρθηκε ε, το εμβόλιο για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, HPV. Αυτά πώς θα ρυθμίζετε τα θέματα για να ξέρουμε πραγματικά τι τρέχει. Γιατί τώρα μόνο ασφάλεια δημιουργούμε μεταξύ των ασθενών και των γονέων, αν θα πρέπει να εμβολιάσουν τα κορίτσια τους κτλ. Ε, αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά ε, ευρύτερο. Δεν είναι μόνο για τον ιό των θυλωμάτων HPV. Κάτι άλλο που ανέφερε η κυρία Κονέτσνα έχει να κάνει με την ε, επαναχρησιμοποίηση κάποιων φαρμάκων που ε, κυκλοφορούν ε, ελεύθερα, το, τα οποία ξαναπατεντάρονται. 380 ευρώ πουλάνε τώρα με το ιδιοσκεύασμα ποντέβαν τη, τη μάρκα και είναι ε, ή μια άλλη ουσία που πωλείται 210 ευρώ ένα σκεύασμα, όχι, διορθώνει ο 180 για ένα μήνα, αλλά 12.100 όταν χρησιμοποιείτε για α, άλλους σκοπούς γονιμότητας. ή ε, θέματα υπέρτασης. Δεν χρειάζεται να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωση στους γιατρούς. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ γνωστά, είναι ενώσιμα και τα λοιπά και κυκλοφορούν ελεύθερα. Και κάτι άλλο για την προσαρμογή ε, και τα μονοπάτια προσαρμογής. Adaptive Pathways. Είναι μια ε, ευρεσιτεχνία δικιά σας, συμμετέχουν και ΜΚΟ και άλλοι, αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Μόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις να παρακάμπτεται αυτή η διαδικασία και να υπάρχουν αυτές οι ταχείες fast track. Και μετά να υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε ασθενεί. Όλοι γνωρίζουμε ασθενεί που κλαίνε για να υπάρξει νέο φάρμακο. Αλλά έρχεται ένα φάρμακο που δεν ξέρουμε τι έχει, παρενέργειε, ανεπιθύμητε ενέργειε. Σοκαρίστηκα όταν το άκουσα αυτό για πρώτη φορά. Βεβαίω, σε ιδιαίτερα έκτακτε και σπάνιε περιπτώσει, ναι, αλλά να το έχετε τώρα και μοντέλο. Αυτά όλα είναι στην νομοθεσία. Ε, τα προβλέπει ω απόλυτε εξαιρέσει θα πρέπει να μας διαβεβαίωσετε ότι δεν πρόκειται να είναι ένας τρόπος λειτουργίας φυσιολογικός. Τα έχω δει και τα λέω αυτά και στις τηλεοράσεις και ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Θα πρέπει να προστατεύουμε και το φάρμακο και τη δράση του και τις γνώσεις που έχουμε σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, καθηγητή Ράζη που είναι εδώ μαζί μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τον ε, συγχαρώ για τις πρόσφατες προσπάθειές του, για, τις, ε, για την αύξηση της διαφάνειας για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές και την απαραίτητη ενθάρρυνση και προς τις ρυθμιστικές αρχές. Θα ήθελα να πεντρωθώ σε ένα σημείο τακτική χρήση συγκεκριμένων αντιβιωτικών που θα πρέπει να, ε, στα ζώα που θα πρέπει να απαγορευτεί. Όμως τα δεδομένα του ΕΟΦ από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι υπάρχει υπερβολική χρήση ισχυρών ε, αντιβιωτικών και αυτό είναι σημαντικός παράγοντας στην ε, αύξηση της αντοχής στα αντιβιωτικά. είναι κάτι το οποίο ε, θέτει σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υγεία γιατί αυξάνει την αντιμικροβιακή αντοχή ακόμα και στα πλέον ε, ισχυρά φάρμακα. Ποιε ε, είναι οι δικέ σα απόψει προ αυτό. Θεωρείτε ότι αυτή η αξιμένη χρήση επιβεβαιώνει ότι αυτή η ε, ήπια και προαιρετική προσέγγιση δεν λειτουργεί πλέον και θα πρέπει να, ε, πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη διαφορετική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαστε που σας βλέπουμε στην Επιτροπή μας σήμερα Έχουμε όλοι ερωτήσεις προφανώς. Πρώτη ερώτηση και ένα σχόλιο μαζί. Έχει να κάνει με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις για το Brexit και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και συνέπειες για τον ΕΟΦ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ρωτήσω το εξής. θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύετε, μια γρήγορη επικοινωνιακή τακτική ή όχι. Και σε ποια χώρα θα πάτε. Προτιμάτε τα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως και τα καινούρια. Ξέρουμε ότι είναι σε νησί αυτή τη στιγμή ο ΕΟΦ ε, κάπως απομονωμένος στο μέλλον δεν θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάτι πιο κεντρικό. Πώς το βλέπετε αυτό. Δεύτερον, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οδηγία του 2011, 62 2011, να εφαρμόζεται σωστά. Αυτή η οδηγία αφορά τα πλαστά και τις απομιμήσεις φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην κυκλοφορούν. Ε, και τέθηκε σε ισχύ στις 2 πρώτου 2013 παντού. Και φαρμακοεπαγρύπνηση ε, θα πρέπει να ήταν εξασφαλισμένη μέχρι τις 2 πρώτου 2017. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, οπότε φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια κατεξοδότηση πράξη ε, που παρέτεινε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου του 2017 ε, την προθεσμία αυτή. Έχουμε όμως Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Από πού και ως που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει όλα αυτά να τα διεκπαιρεώσει με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Αναθέτει στη φαρμακοβιομηχανία κάποια πράγματα που είναι δική σας αρμοδιότητα. Και τι κάνετε εσείς, πώς συμμετέχετε σε αυτό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι κατεξοχήν αρμόδιος για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, για την υγεία ε, και τα λοιπά και για το φάρμακο. Και έχουμε προβλήματα γενικότερα τώρα για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο, το Ευρωπαϊκό Hub. Όλα αυτά έρχονται πολύ αργά και δεν αποδίδουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπορντ, εκπρόσωπο το, πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ μετά από μια μικρή ανάπαυλα. Για το Brexit, αν θεωρήσουμε ότι θα ε, ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 50 το Μάρτιο, έστω ότι συμβεί αυτό, με ένα ε, χρονικό πλαίσιο δύο ετών. Ξέρω ότι δεν είναι απόφαση του ΕΟΦ, αλλά αυτό μας δίνει ένα μικρό χρονικό περιθώριο. Νομίζω θα πρέπει να ασκηθεί η πίεση στο Συμβούλιο για να λάβει απόφαση. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν όταν συμβεί όντως το Brexit να είναι άλλη μία μέρα όπως όλες οι άλλες για τον ΕΟΦ να υπάρξει ε, μετακαταστασή του και μια πολύ ομαλή μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει μια ομάδα που ασχολείται ακριβώς με αυτό στον ΕΟΦ. Όχι μόνο ε, για το κλίμα που επικρατεί, ένα κλίμα ανησυχία όπως αναφέρατε, αλλά και μια ομάδα που θα διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν ε, όπως πρέπει. Γιατί υπάρχουν ε, τόσοι μνηστήρες, αν θέλετε, που θέλουν να φιλοξενήσουν τον ΕΟΦΕ στην πόλη τους, που θα πρέπει να δούμε ότι όλα θα γίνουν καλά. Μετά, ο εκτελεστικός διευθυντής, σε πολύ ωραία και όμορφα αναφέρθηκε στους, ε, στους περιορισμούς ως προς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, σε, σε ποιον κλάδο θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Εγώ από την εμπειρία μου ως πολιτικού και επιτρόπου δεν γνωρίζω κανένα θεσμικό όργανο που να λέει ότι έχει πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι λένε ότι τους λείπει κόσμος και προσωπικό. Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα με παράδειγμα με το να λέμε ε, για τις ανάγκες που θα υπάρχουν κάποια στιγμή ε, λόγω της μετεκατάστασης. Δεύτερον, με καλύτερη αναδιοργάνωση για αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων που έχετε ήδη στη διάθεσή σας. Ποιες είναι οι σκέψεις σας ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταίο σχόλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ρουίζ. Παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω, μόνο μία γενική παρατήρηση η συνεργασία μας ε, με τον ε, καθηγητή Ράση και το επιτελείο του είναι εξαιρετική. Κάθε μέρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτές ε, τις σχέσεις, αυτή τη συνεργασία, όχι μόνο όταν συναντιόμαστε και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, αλλά καθημερινά συνεργαζόμαστε σε μία σειρά project και για την έγκριση φαρμάκων, αλλά και για, την, ε, και για νέες πρωτοβουλίες σε διεθνές ε, επίπεδο. Ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να τον ευχαριστήσω και προσβλέπω σε περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον. Βεβαίως και δεδομένου του Brexit θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο και πάλι λοιπόν στον κύριο Ράση για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να θυμηθώ όλα τα σχολιά σας. Αν ξεχάσω κάτι, παρακαλώ υπήρχε το μου. Λοιπόν, πολλοί από σας αναφερθήκατε στο Brexit. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω συνολικά. Κάποιος ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημα ήδη τώρα πριν από το Brexit. Πολύ καλό ερώτημα. Υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας. Αυτό ανέφερα προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι ε, και το προσωπικό μας έχει χάσει λίγο το κίνητρό του, αν θέλετε. Και εξετάζουμε επιπλέον μέτρα για να στηρίξουμε το προσωπικό μας έχουμε αρχίσει και το κυνήγι κεφαλών εντό αγωγικών. Κάποιοι σκέφτονται ήδη να φύγουν, δεν ξέρουν κατά πόσο ε, πρέπει να πάρουν το ρίσκο και να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή πρέπει να φύγουν. Ήδη έξι μέλη μας ε, ε, υπέβαλαν την παρέτησή τους το τελευταίο εξάμενο, είχαμε πολύ λιγότερες το τελευταία πέντε έτη. Παρακολουθούμε την τάση για τη διαδικασία επιλογής ε, προσωπικού που έχουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι πολύ καλοί υποψήφοι αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Θέλουμε να δούμε αν συνδέεται αυτό ή όχι. Αυτά συμβαίνουν ήδη πριν από ένα πιθανό Brexit. Ένα μέτρο μετριασμού είναι ε, η συνεχής επικαιροποίηση, και του φόρτου εργασίας. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο υπάρχει πλεονάζον δυναμικό ε, στο κράτος μέλος για να αναλάβει το 20% του φόρτου εργασίας που καλύπτει αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να ενισχύσουμε το δυναμικό αυτό έχουμε θεσπίσει ένα κέντρο ε, για να καταρτήσουμε εμπειρογνώμονες ανά την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ απλό αλλά και πολύ αποτελεσματικό μοντέλο. Ουσιαστικά παρέχουμε στήριξη και στον καταρτιστή, εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο, ε, όπου και αν αυτοί βρίσκονται στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Ο κύριος Βόρκ ρώτησε κατά πόσο υπάρχει μια ειδική ομάδα. Υπάρχει μια ειδική ομάδα λοιπόν που έχει αναλάβει όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα πώς θα γίνει η επανακατάστασή μας. Δεν μας απασχολεί τόσο το τεχνικό σκέλος. Μόλις πριν από δύο χρόνια μεταφερθήκαμε σε νέο κτίριο, μόλις μία ώρα σταματήσαμε τις εργασίες μας. Επομένως είμαστε εκπαιδευμένοι. Βεβαίω το να αλλάξουμε χώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μας απασχολεί τόσο λοιπόν το θέμα της ε, όσο ε, το θέμα της ε, λειτουργίας μας, της συνδεσιμότητας. 40.000 εμπειρογνώμονες κάθε χρόνο συνεργάζονται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αεροδρόμιο, χρειαζόμαστε ε, επίγειες ε, μεταφορές, 250 δωμάτια ε, ε αναβράδυ, 5 βράδια την εβδομάδα. Υπάρχουν τέτοιες τεχνικές δυσκολίες. Κάποιος άλλος ε, ρώτησε ποια είναι η δική μας επιρροή. Μηδενική είναι η επιρροή μας. Δεν έχουμε κανέναν ρόλο για το πού θα πάμε. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε δηλαδή αυτή την απόφαση. Από ό,τι ξέρω, αυτό εναπόκειται πλήρως ε, στο Συμβούλιο, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, πόσο ζωτική σημασία είναι η ασφάλεια ε, και η δημόσια υγεία ε, των Ευρωπαίων πολιτών και πώς όλα αυτά κινδυνεύουν αν ε, διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΦ. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που αφορούσαν τον Brexit. Αλλιώς μπορώ να επανέλθω. Με τα χαράς. Ε, για την αναθεώρηση για το εμβόλιο για τον HPV. Έχετε δίκιο. Η Επιτροπή μας εξέτασε, εξέτασε συγγνώμη, ε, όλα τα επιστημονικά δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο σύνδρομα που αναφέρατε προηγουμένως έχουν την ίδια συχνότητα και στον πληθυσμό που έχει δεχτεί το εμβόλιο και στον πληθυσμό που δεν το έχει λάβει. Επομένω δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και των δύο συνδρόμων, τουλάχιστον με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε, αν υπάρξει διαφωνία από αυτού, ελπίζουμε λοιπόν αυτοί που διαφωνούν να προσκομίσουν και τα στοιχεία, αντί απλώς να προσπαθούν ε, να διαψεύσουν ε, τα θεσμικά όργανα. Εμείς ακολουθούμε τα επιστημονικά δεδομένα. Αν υπάρξουν νέα επιστημονικά δεδομένα, όπως πάντα, ε, θα αποφανθούμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Το ίδιο, και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνατε να το ε, επισημάνω, το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τον αυτισμό. Όλοι ξέρουμε πλέον ότι τα εμβόλια και ο αυτισμός δεν ε, στέμνονται κάπως, δεν προκαλεί το ένα το άλλο. Υπήρξε λοιπόν μία ψευδής ε, ιστορία για ορισμένα κρούσματα. Τα δύο αυτά θέματα όμως ε, είναι ζητήματα μυθοπλασίας και μόνο, που έχουν προκύψει από τον τύπο. Πώς ε, ε, για την ανάκληση της ε, θέσης εμπορία υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες, ε, μπορεί να γίνει και από ένα πρόσωπο. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για να δούμε κατά πόσο πρέπει να υπάρξει ανάκληση ή όχι. ή αν θα πρέπει να διευκρινίσουν χωρίς ανάκληση. Έτσι έχει διαδικασία. για την ε, προσέγγιση μη εμβολιακή, εμβολιαστική. Είναι κάτι το οποίο μας ε, προβληματίζει ιδιαίτερος. Βέβαια, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να κάνουν εκστρατείε για να προωθήσουν τον εμβολιασμό, όμως μας προβληματίζει ιδιαίτερα αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ε, ελπίζουμε να υπάρξει μία εκστρατεία. Έχουμε λάβει μεγάλη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ε, της, των πρωτοβουλίων για την αντιμικροβιακή αντοχή. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε αυτή την, ε, το, ντροπιαστικό φαινόμενο να έχουμε θανάτους από ασθένειες όπως η λαρά. εξαιτία ε, του μη εμβολιασμού του πληθυσμού μα. Επομένω, μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε ενεργά ε, να κάνουμε εκστρατεία. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αναλάβει. Για αυτό το adaptive Pathways. Νομίζω ότι πολλοί από εσά ε, το αναφέρατε. Πρώτα θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Υπήρχε αίτηση για 62 φάρμακα για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα ε, των προσαρμοστικών διόδων. Εξετάσαμε μόνο 18 και μόλις 7 εγκρίθηκαν. Επιτρέψαμε δηλαδή να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι ίσως επιτυχής η διαδικασία, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι διευκολύνουμε την πρόσβαση στην αγορά. Τι σημαίνει το να ενταχθεί κανείς σε αυτό το πρόγραμμα. Ουσιαστικά θέλουμε να καλύψουμε μια ιατρική ανάγκη που επήγει και δεν έχει ακόμα καλυφθεί και υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, αλλά βλέπουμε ότι είναι αδύνατον να καταλήξουμε σε εύρο στα επιστημονικά στοιχεία με τον παραδοσιακό τρόπο. Μιλούμε για μικρούς πληθυσμούς, εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες, όπου ε, μία παραδοσιακή τυχεοποιημένη επιστημονική μελέτη δεν μπορεί να διεξαχθεί ή θα πάρει υπερβολικά πολύ χρόνο ή ο σχεδιασμός της μελέτης θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στην ε, πραγματικότητα της ασθένειας την οποία μελετούμε. Η μεθοδολογία ε, κινδύνου ωφέλους δεν έχει αλλάξει. Επομένω, αν θεωρήσουμε ότι εδώ θέλουμε να καλύψουμε έναν πολύ μικρό πληθυσμό, όπου είναι ξεκάθαρη η ιατρική ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί, εκεί η σχέση ωφέλεια κινδύνου είναι μεγαλύτερη, όχι μικρότερη. Η αβεβαιότητα είναι μικρότερη, όχι υψηλότερη. Το πρόβλημα είναι λοιπόν που στο τελευταίο τμήμα της αλυσίδας, στο τελευταίο κρίκο, πώς διασφαλίζουμε ότι η συνταγογράφηση ακολουθεί τους κανόνες και ούτω καθεξής. Αυτά τα ζητήματα δεν έχουν επιληθεί. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα το Adaptive Pathways. Είναι μια διαδικασία προβληματισμού, μια προσέγγιση ε, που ε, ενέχει πολλά σημεία που εκκρεμούν και θα πρέπει να συζητηθούν και να επιληθούν. Είναι μια πιθανή προσέγγιση για ε, ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί. Στις 8 Οκτωβρίου με τα χαράς μπορώ να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ε, συνάντηση μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκρινίσουμε όλες αυτές τις πτυχές, να δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε με αυτή την, ε, σε αυτή την οδό στο μέλλον, τι πρέπει να αλλάξει, να βελτιωθεί και ελπίζουμε με την συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αν υπάρχουν καλύτερες λύσεις, ε, να τις βρούμε ή να βελτιώσουμε αυτή τη λύση που έχουμε βρει εμείς. Ωστόσο, προς το παρόν δεν βλέπω πολλές νέες προτάσεις. για να έχουμε αυτά τα επιστημονικά στοιχεία χωρίς να σχεδιάσουμε την ε, ε, επανεξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων και των σχεδιασμών νέων μελετών όταν είναι πολύ δύσκολο να ε, παράξουμε αυτά τα δεδομένα. Άλλο πρόβλημα. Για τις ευρεσιτεχνίες. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε και ε, για την επέκταση των ευρεσιτεχνιών, για το κοστολόγιο, για το τρόπο με τον οποίο Κάποιοι προσπαθούν να επωφεληθούν, να κερδοσκοπήσουν ε, για λόγους εμπορικούς παρά να ανταποκριθούν σε κάποια ιατρική ανάγκη. για την κανονική ας πούμε πρόσβαση στην αγορά. Φοβάμαι ότι αυτό είναι τελείως εκτός της δικής μας εντολής και αρμοδιότητας. Θέματα ευρεσιτεχνιών δεν έχουμε καθόλου αρμοδιότητα μόνο για κάποια παιδιατρικά. Τι άλλο με ρωτήσατε. Α, την πρόσβαση. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Οι ελλείψεις, οι τεχνητές και οι παράλληλες εισαγωγές. Και πάλι, εμείς δεν μπορούμε παρά ε, να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις που έχουν να κάνουν με θέματα ποιότητας. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε στο HNA που είναι δηλαδή ε, εκπροσωπούνται όλοι οι εθνικοί οργανισμοί φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, δούμε αυτό το πρόβλημα. Οι παράλληλες εισαγωγές, εξαγωγές, τεχνητές ελλείψεις και αυτά δεν είναι κάτι το οποίο τις δικές μας αρμοδιότητες για να παρέμβουμε εμείς. Αυτό είναι εκτός της αρμοδιότητας και της εντολής μας. Και μάλιστα είναι και σε άλλη γενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κάνει στη δικιά μας. Είναι μέγα πρόβλημα, δεν διαφωνώ και θα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητούμε, έχει φτάσει η ώρα και γιατί έχει συνέπειε. σύγκρουση συμφερόντων των ε, εμπειρογνωμόνων μας. Αυτό μπορεί να το δει κανείς με δύο τρόπους. Μονίμως έχουμε έξι ε, ε, εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που ελέγχουν όλη την υπηρεσία μας, όλο το δίκτυο και παρακολουθούν και ελέγχουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Ε, γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, γίνονται εκ των υστέρων έλεγχοι και τυχαίοι έλεγχοι. Νομίζω ότι έχουμε την πιο αυστηρή πολιτική σύγκρουση συμφερόντων παγκοσμίω. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια αυτό. Χωρίς να είμαστε <laughs> αστυνομικό σώμα. Οι καταγγέλλοντες είναι ευπρόσδεκτοι, whistleblowers και όποιο γνωρίζει οτιδήποτε έρχεται να μας το καταγγείλει, το ελέγχουμε. Αλλά πολύ πιο πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε δυστυχώς. Η πολιτική μας για τη σύγκρουση συμφερόντων νομίζω είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί αυτό τον καιρό στην νομοθεσία. Η νομοθεσία και πάλι είναι πέραν των αρμοδιοτήτων μας. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα. Well, I, I think we have three policies. Έχουμε τρεις πολιτικές για τρία επίπεδα, Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και μια διαδικασία ε, απιστίας. Ε, όλα αυτά τα δημοσιεύουμε. Και ε, όποιος εξωτερικός γνωρίζει οτιδήποτε, με χαρά να μας το... Ε, μεταβιβάσει, να μας το διαβάσει και θα δράσουμε. Τι άλλο. Α, για την ε, χρήση ρουτίνας των αντιβιωτικών που έχουμε. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε κατά 65% ε, τα αντιβιωτικά, τα κτηνιατρικά η χολιστίνη, η χολιστίνη 65% Η έκτη έκθεση μας έδειξε ότι υπάρχει μία μείωση των ε, αντιβιωτικών στην ε, κτηνοτροφία. Βέβαια, όντως, ε, είναι μεγάλο το ποσοστό ακόμα, ξέρω ότι στην Κομισιόν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση στην νομοθεσία. Εμείς θέλουμε, θέλουμε η νομοθεσία αυτή της Κομισιόν να προχωρήσει και να επιβάλλουμε μείωση της, της περιτής χρήσης των αντιβιωτικών στην, ε, τροφία ή για τα ζώα γενικότερα. Βέβαια για, για, για τη συνανθρώπινη πλευρά το μεγάλο πρόβλημα είναι η ε, κακή χρήση των ε, αντιβιωτικών που τα παίρνουν χωρίς συνταγή παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ουσιαστικό που αντιμετωπίζουμε και υπάρχει μια δράση σημαντική την οποία έχει ξεκινήσει η Κομισιόν και στην οποία να συμμετέχουμε ε, σε συντονισμό με, τις άλλες, με τις δύο οργανισμούς, το CBC και, την, ε, και ε, το EFSI βέβαια. Α, τα πλαστά τώρα. Υπάρχει ένα ε, πολύ ε, σοβαρό πρόβλημα, τα πλαστά φάρμακα. Αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, μπορούμε να κάνουμε δημοσιεύσεις. Άμεση παρέμβαση δεν μπορούμε να κάνουμε. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να δοθεί μια απάντηση, που είναι το εξής. Εάν είμαστε, αν είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν πλαστά, τέλος πάντων, παραποιημένα φάρμακα στην Ευρώπη. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Βέβαια, η Ευρώπη είναι ικανή να ε, περιορίσει το πρόβλημα αυτό, τις απομιμήσεις ε, στα φάρμακα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ε, τα websites που κυκλοφορούν, διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φαρμάκων που εμφανίζονται στα διάφορα websites, διάφορους τοπούς, είναι απομιμήσεις. Τώρα, τι γίνεται όταν στις χώρες που λειτουργεί το παραδοσιακό σύστημα των φαρμάκων, ε, εκεί το ποσοστό των απομιμήσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εμείς συνεισφέρουμε να τον περισσότερο σε αυτή την προσέγγιση ότι ε, λέμε ότι Όταν έχουμε το φάρμακο ε, σε μια, σε, σε μια συγκεκριμένη συσκευασία, ορίζεται η τιμή. Βέβαια, μιλάμε για ποινικέ ε, ενέργειες, ε, ελέγχουμε αυτή την προσέγγιση από που εφαρμόζουν κάποιοι. Ξέρω ότι στα τελωνία και στις, ε, στις γίνεται ο έλεγχο σε κάποια κράτη-μέλη, στους μεθοριακούς ε, σταθμούς. Θα δούμε τι θα γίνει. Η τιμή, η κοστολόγηση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό μεν, αλλά δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική για να ελαφρύνουμε το φορτίο, αν θέλετε, της έρευνας. Ε, γι' αυτό βέβαια για τις επιχειρήσεις μεταφράζεται όσο όφελος ε, στην αγορά. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με το HB, ε, τα, τα σώματα αυτά, έτσι ώστε να υπολογίσουμε σωστά την ε, προστιθέμενη αξία των νέων φαρμάκων. Τώρα βέβαια πώς αυτή η προστιθέμενη αξία θα ε, μεταφερθεί και θα ερμηνευθεί στην τιμή του φαρμάκου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, διότι ε, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει κατά πολύ στα κράτη-μέλη. Περιορισμός των πόρων. Έχουμε περιορισμούς των πόρων και θα σας ε, δώσω κάποια στοιχεία. Οι περισσότεροι λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους και όλοι οι διευθυντές, ας πούμε, και σε μένα έρχονται και μου λένε χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Αυτή είναι μία φυσιολογική προσέγγιση. Όμως, εφόσον έχεις ε, εφαρμόσει τρεις κανονισμούς χωρίς σημαντική ε, βελτίωση ε, στον αριθμό του προσωπικού, ε, τότε το πρόβλημα γίνεται σημαντικό. Μπορούμε να δώσουμε κάποια, κάποιες θέσεις που αφορούν όχι τόσο ευαίσθητες ευαίσθητους τομείς, ε, αλλά σε ευαίσθητους τομείς χρειαζόμαστε ε, πολύ έμπειρους επαγγελματίες. Για την πρόσβαση στην αγορά έχουμε, ε, η πρόσβαση στα έγγραφα έχουν 25 άτομα μόνο. Δηλαδή, εφόσον είναι 25 πρέπει να είναι οι καλύτεροι εξημών. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά καλύτερα, που μπορούν να χειριστούν τα επιστημονικά δεδομένα και αυτό ήταν εις βάρος βέβαια των βασικών μας δραστηριοτήτων. Όταν ξεκινήσαμε κάποιες δραστηριότητες ε, προσπαθούμε να ε, βελτιώσουμε κάποιους ε, οργανισμούς, κάποιους νέους επιχειρηματι... κάποιες νέες επιχειρήσεις τέλος πάντων, κάποιες νέες εταιρείες οι οποίοι οι οποίες ε, ε, έχουν μεν ε, καλές ιδέες, έχουν καλούς επιστήμονες, έχουν μία αποτελεσματική μέθοδος, όμως κάποια διαδικασία, οι διαδικασίες που εφαρμόζουν λόγω απειρίας δεν είναι σωστές και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και, την, και τον ασθενή. Επομένως, αυτό το οποίο θέλουμε να, να κάνουμε είναι να δώσουμε, να δώσουμε, να παρέχουμε τη βοήθεια που χρειάζεται. Δώσαμε 600, στο τελευταίο χρόνο 600 ε, επιστημονικές συμβουλές. Ε, και επίσης ε, μας είπαν ότι έπρεπε να μειώσουμε κατά 2% κάθε χρόνο την, το εργατικό μας δυναμικό. Ενώ αντίθετα χρειάζεται να, αυξήσουμε. Βέβαια, την αύξηση είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί. Ο προϋπολογισμός μας είναι πολύ καλός, είναι θετικός ε, και το έχουμε εξηγήσει αυτό. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστούν ε, ε, και σε μας επιχειρηματικές πρακτικές, γιατί όντως πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα βέβαια να πω τα κακά ε, σε αυτή την επιτροπή δεν πρέπει γιατί ε, μας έρχεται υποστηρίξει πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάτι. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ αυτό το σημείο και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ράζη για, αυτή την, για αυτές τις τόσο λεπτομερείς εξηγήσει που μας έδωσε και για τις ε, απαντήσεις του. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι ένα σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για τον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα. Και θα δώσω τον λόγο ε, κατευθείαν στους συνεισηγητές, ξεκινώντας από την κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για ένα ψήφισμα που αφορά τον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα αυτό το ψήφισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Καταρχάς διότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση προς την Κομισιό που στις αρχές του 2017 θα πρέπει να υποβάλει μία έκθεση για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του παιδιατρικού κανονισμού που υπάρχει από το 2006. Λόγω της μεγάλης ζήτησης από πλευράς των παιδιάτρων και των ενώσεων των γονέων, γονέων ασθενών ε, άρρωστων παιδιών θα πρέπει η έκθεση αυτή να, να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ασκήσει πιέσεις εδώ και καιρό Δυστυχώς όμως ε, έπρεπε να περιμένουμε στις αρχές, αρχές του 2017. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να μπορούμε να πούμε στην Κομισιόν συγκεκριμένα εν ώψη της δημοσίευσης αυτής της έκθεσης ποιες είναι οι, οι τομείς αλλαγής, αλλαγών ε, που θα θέλαμε, οι τροπολογιών που θα θέλαμε να προτείνουμε. Ήμουνα εισηγήτρια στον κανονισμό του 2006. Το κείμενο αυτό επέτρεψε να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι, κυρίως κυρίως ε, υποχρεώνοντας ε, τα εργαστήρια να κάνουν ε, και τις έρευνες για τις συνέπειες προς τα παιδιά όλων των φαρμάκων τα οποία προορίζονται για ενήλικες, όμως σε, κάποιες, για σε κάποιους τομείς ιατρικούς και στον τομέα του καρκίνου των παιδιών, ο κανονισμός αυτός έχει περιοριστεί. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι επίγονο να προωθηθεί αυτός ο κανονισμός για τα παιδιατρικά φάρμακα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να ε, υπάρχει μια πλήρης αναθεώρηση του κανονισμού, εκτός βέβαια αν η Κομισιόν θεωρήσει ε, μέσα από την έκθεσή, του, την έκθεσή της ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσει την κατάσταση. Εγώ λέω ότι είναι επίγον να γίνει η αναθεώρηση, βέβαια πλήρης αναθεώρηση χρειάζεται πολύ χρόνο και οι ασθενεί δεν έχουν χρόνο, δεν μπορούν να περιμένουν. Επίσης το κείμενο ως έχει θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή βάση εργασίας, μπορεί όμως να γίνει και θα μπορούσε να είναι όμως αντιπαραγωγικό αν αμφισβητήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του. Όμως μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές μέσω κανονιστικών διαδικασίων και μέσω κατευθυντηρίων γραμμών της, ε, του οργανισμού και θα δώσω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη η υποχρέωση ε, των ε, ερευνών για τα παιδιατρικά φάρμακα, ε, όχι μόνο πάνω στο φάρμακο, αλλά πάνω στο μόριο το οποίο έχει βρεθεί για τους ενήλικες και χρησιμοποιείται για βάση των φαρμάκων για τους ενήλικες. Διότι μέχρι στιγμής δεν γίνονται αυτές οι έρευνες γιατί χρησιμοποιείται η πρόφαση ότι ε, η ασθένεια αυτή δεν υπάρχει για τα παιδιά. Όχι, εμείς ε, θέλουμε να περιορίσουμε τον τόπο περισσότερο τις εξαιρέσεις, διότι έχουμε επιτρέψει πάρα πολλές εξαιρέσεις και δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεύτερον, θα πρέπει τα ε, παιδιατρικά σχέδια έρευνας θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα και θα πρέπει να επιτραπεί ο διάλογος, αν θέλετε, ανάμεσα στα εργαστήρια και στην ε, και στον οργανισμό. Τα παιδιοτρικά σχέδια αυτή τη στιγμή είτε εγκαταλείπονται είτε καθυστερούν λόγω μη αξιόπιστων ε, ε, πληροφοριών. Πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι αλλά πιο συστηματικοί. Και τελευταίο σημείο θα πρέπει να επανα... επανεξετάσουμε, να αναθεωρήσουμε το όλο σύστημα για να δούμε πόσο μπορούμε να, πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά. Έχουμε κίνητρα αυτή τη στιγμή, έχουμε έξι μήνες πραγματικούς για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα μέτρα αυτά όμως ε, έρχονται πάρα πολύ αργά στην όλη διαδικασία και δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Επίσης δεν υπάρχει και κανένα κίνητρο για τις, για τις παιδιατρικές ενδείξεις. Επομένως οι έξι μήνες προστασίας είναι χρήσιμοι όταν ένα φάρμακο κυκλοφορεί στο εμπόριο και για τους ενήλικες και για τα παιδιά, όμως δεν ε, χρησιμεύουν εάν πρόκειται για μία παιδιατρική μόνο ένδειξη, διότι στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ενδείξεις που είναι σπάνιες, αλλά για αγορές που είναι πολύ περιορισμένες. Επομένως, εάν βελτιώσουμε τα κίνητρα, Ταυτόχρονα μπορούμε να επιβάλλουμε και αποτελεσματικές κυρώσεις για τα εργαστήρια τα οποία δεν θα σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Και με τον τρόπο αυτό που ο διατρικός κανονισμός θα γίνει πιο χρήσιμος και αποτελεσματικός. Επομένως, γιατί λέω τώρα ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μια πλήρη αναθεώρηση αλλά θα έπρεπε να έχουμε μερική αναθεώρηση. Γιατί τα μέτρα αυτά ήδη υπάρχουν στον κανονισμό, τα οποία ανέφερα, υπάρχουν ήδη στον κανονισμό και μπορούν απλώς να εφαρμοστούν γρήγορα, ε, εάν και εφόσον υπάρχει μια διακομματική ε, υποστήριξη και το συζήτησα με τους συναδέλφους, ε, πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να δράσουμε από κοινού προς τον σκοπό αυτό, προς όφελος και προς το συμφέρον των άρρωστων παιδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη έχουμε υπογραμμίσει το, την σημασία αυτής της συζήτησης. Ε, απόλυτα τις ε, προθέσεις που παρουσίασε η συνάδελφος, ότι θα πρέπει δηλαδή να δράσουμε γρήγορα γιατί πρόκειται για ένα θέμα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ανεξάρτητα από τα περιστατικά τοπία και τους αριθμούς που γνωρίζουμε, 6.000 ασθενείς, ε, παιδιά ή ενήλικες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Και πέραν αυτού, αυτών των αριθμών βαρύνει και στη σκέψη μας και ο αριθμός των ασθενών που επιβίωσαν μένα αλλά έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες ε, στην ε, ποιότητα ζωής τους λόγω της ασθένειας. Και πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να επανεξεταστεί βγάζοντας, αφαιρώντας κάποιες ε, αντιφάσεις ε, κάποια, σε κάποια σημεία ασαφή. Κυρίως όσον αφορά την αξιοποίηση του μηχανισμού δράσης. Δηλαδή και να μην μιλάμε για προληπτική χρήση των, φα... ογκολογικών φαρμάκων στην ε, ενήλικη, της ενήλικης, ε, των ενηλίκων. Γιατί όπως ξέρουμε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολλές και καλές. Και είναι αρκετά δύσκολο, για να μην πω και αδύνατον, ένας όγκος, ένας καρκινικός όγκος ε, των ενηλίκων να, εμφαρμοστεί και στα παιδιά, να εμφανιστεί και στα παιδιά. Όμως κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στους ενήλικες έχουν ε, αποτελεσματικότητα και στα παιδιά σε σχέση με ε, όγκους που πολύ συχνά εμφανίζονται στα παιδιά και όχι στους ενήλικες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μπέρδεμα εδώ, υπάρχει το, ένα θέμα για τα κίνητρα, τα οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Τα κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε στην έρευνα για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά που ενδεχόμενα ε, μπορεί τα φάρμακα αυτά να χρησιμοποιούνται σπάνια μεν για τα παιδιά, όμως η κοινωνική τους προστιθέμενη αξία είναι τεράστια. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ε, ένα σημείο συμφωνίας όσον αφορά τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και να δημιουργηθούν και δίκτυα ενδιαφέροντος και δίκτυα έρευνας, δηλαδή να συμμετέχουν και δημόσια εργαστήρια ερευνητικά, ε, πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια. Νομίζω ότι και αυτοί μπορούν να εμπλακούν στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιέκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα που εξετάζουμε σήμερα για τα παιδιατρικά φάρμακα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Γιατί υπάρχει ανάγκη να στρέψουμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια πήγουσα ανάγκη αναθεώρησης ε, του κανονισμού 1902-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Είναι ευρέως γνωστός ως ο παιδιατρικός κανονισμός πλέον έχουν περάσει 10 χρόνια από την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού, 10 χρόνια για την ιατρική, ιδίω ε, με βάση τις ε, σύγχρονες τεχνολογίες, είναι μια ολόκληρη εποχή. Αλλάζουν λοιπόν ραγδαία και οι θεραπείες, οι ιατροί χρησιμοποιούν ε, τεχνολογίες εχμής στον εξοπλισμό τους, με εξατομικευμένες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία ε, αντίστοιχη τροποποίηση της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε μια αντιστοιχη τροποποιηση της νομοθεσιας χρειαζομαστε μια εκθεση που θα υποβληθεί στα τέλη της χρονιάς ή ε, στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Χρειαζόμαστε λοιπόν και έναν στόχο βελτίωσης ε, του κανονισμού αυτού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, με τη δημόσια υγεία και πιο συγκεκριμένα με την υγεία των παιδιών. Ο σκοπός λοιπόν της αναθεώρησης αυτού του κανονισμού θα πρέπει αφενός να είναι προσβασιμότητα και με προσβασιμότητα εννοώ και προσιτές τιμές, ε, προσιτό κόστος θεραπείας για τις ε, τεχνολογίες εχμής. Από την άλλη όμως θα πρέπει και να ενθαρρύνουμε τις φαρμακοβιομηχανίες και όλους όσοι ασχολούνται ακριβώς με την ε, φαρμακευτική έρευνα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα που αναφέραμε και προηγουμένω. Πολύ συχνά όταν μιλούμε για το δίκαιο ευρεσιτεχνιών υπάρχουν εντάσει σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία για τα φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο ε, να μειώσουμε αυτές τις ε, εντάσεις να ευθυγραμμίζονται περισσότερο οι δαπάνες ε, στα πρώιμα στάδια των ερευνών των φαρμακοβιομηχανών φαρμακοβιομηχανιών από τη μία και του προπολογισμού των κρατών μελών από την άλλη. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις ε, διαθέσιμες μεθόδους για τη διασφάλιση της δημόσιας Το θέμα εδώ είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που πάσουν από ογκολογικές ασθένειες, αλλά και άλλες πολύ σπάνιες νόσους, που εντοπίζουμε μόνο στα παιδιά και ε, σε πολύ μικρό ποσοστό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο. Ο νέος, οι νέοι κανονισμοί θα βοηθήσουν για να βρούμε νέες, πιο ευέλικτες λύσεις. Για να διαμορφώσουμε μια νέα βάση καλύτερης αξιοποίησης του προπολογισμού των κρατών μελών για την ε, δημόσια υγεία και για την καλύτερη αξιοποίηση των φαρμακευτικών αγωγών για τα παιδιά. Ευχαριστώ κύριο Σπιτιτσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι τα, τα θέματα της, τα, των παιδιατρικών φαρμάκων είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Συμφωνούμε σε, σε γενικές γραμμές με το ψήφισμα αυτό, κυρίως για την έλλειψη ε, φαρμάκων για τις ε, αποκλειστικές παιδιατρικές ε, ασθένειες. Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην Παιδιατρική Επιτροπή. Κυρίως ε, θα ήθελα να πω ότι ε, έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τα κίνητρα γιατί να, ε, που δίνει η, η Κομισιόν σε κάποιες εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, όταν τους δίνουν κάποιες επιδοτήσεις για να κάνουν κάποιες έρευνες σε παιδιατρικά φάρμακα τα, οι επιδοτήσεις γίνονται ακόμα και αν η μια εταιρεία απλά πει ότι κάνει κάποια έρευνα, χωρίς να έχουμε εξακριβώσει ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα ή ασφάλεια. Ε, δηλαδή πολλές φορές ακόμα και η έρευνα για τους ενήλικες μπορεί να επιτρέψει στις φαρμακευτικές εταιρείε απλώς να, παρατεί, να διευρύνουν λίγο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να δείξουν ότι έχουν κάνει και έρευνα για τα, ε, και στην ε, παιδιατρική. Ε, λοιπόν, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα ως έχει, εάν δεν διευκρινιστεί άμεσα το σημείο αυτό. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εγκρίνουμε μία γραμμή που να ευνοεί μόνο ε, τις φαρμακευτικές εταιρείες και ε, όχι την παιδιατρική φροντίδα και θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ρης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω ε, είναι μείζονο σημασία η υγεία των παιδιών, ε, ε, πολύ σημαντικό στόχο πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συζήτηση και επισημαίνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δεύτερη έκθεση ε, για τα παιδιατρικά φάρμακα προς ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι οι κανονισμοί αυτοί έχουν ως στόχο ε, την παροχή των απαραίτητων φαρμάκων προς τα παιδιά για να θεραπεύσουμε αυτές τις ασθένειες. Πρόκειται και για ένα νομοθετικό κίνητρο γιατί συνήθως ε, στρεφόμαστε περισσότερο στις ε, αγορές ε, ενηλίκων. Γι' αυτό, όπως ανέφερε και η κυρία Γκροστέτ, εμείς καταρτήσαμε αυτό τον κανονισμό. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου και τα όσα έλεγαν παλαιότερα η παιδίατροι, ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς μικροί ενήλικες. Και αυτό ήταν και η βάση για αυτούς τους κανονισμούς. Έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και πολύ ε, στοχευμένη παιδιατρική έρευνα. Ο κανονισμός ήταν σίγουρα κάτι που άλλαξε τα πράγματα, Άρδιν, και των λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων. Ε, επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να επηρεάζουν άμεσα την έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, να, να ζητούν συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. Οι κανονισμοί θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ε, τις νέες παιδιατρικές ανάγκες. Επομένω, με βάση ε, της Παιδιατρικής Επιτροπή και του ΕΟΦ, καταλήγουμε στα συμπεράσματά μα. Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί ε, και στα όσα μπορούν να πετύχουν οι κανονισμοί. Οι υποχρεώσει ε, βασίζονται στις εξελίξεις που ε, λαμβάνουν χώρα στον τομέα των φαρμάκων ανηλίκων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο εδώ. Επομένως, η επιπλέον παιδιατρική έρευνα ε, μπορεί να μην ε, καλύπτει νόσους που υπάρχουν μόνο στα παιδιά. Επομένως, εξετάζουμε μεγάλο, με μεγάλη προσοχή τι ακριβώς πρέπει να καλύψουμε. Τα νέα αυτά προϊόντα αντιμετωπίζουν τις ε, πιο διαδεδομένες ε, και επίγουσες ε, παιδιατρικές ανάγκες. Καλύπτουμε λοιπόν τα σημαντικά κενά. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα υποφελούνται νέων ενιών όπως είναι η εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή. ιεραρχούμε ως προτεραιότητα επαρκώς ε, την παιδιατρική έρευνα και έχουμε στοιχεία που να το καταδεικνύουν αυτό. Ταυτόχρονα εξετάζουμε και τον οικονομικό αντίκτυπο των κανονισμών που εστιάζει πιο συγκεκριμένα ε, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης. Είναι δύσκολο λοιπόν το να συλλέξουμε και τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, που κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Σε λίγες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του μηνό αυτού ακόμα Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει μια δημοσία διαβούλευση για να μας δώσουν και ένα feedback ε, οι ενδιαφερόμενοι. Είναι σημαντικό να ακούσουμε ε, όλους τους ενδιαφερομένους πριν ε, τελειώσει, παιδιατρικές επιτροπές, ογκολόγους, βιομηχανία κτλ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να ε, καταλήξει σε συμπεράσματα, ούτε να σας προτείνει ε, δρόμους. Ελπίζουμε μέσα στο 17 να ολοκληρωθεί η έκθεση. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ε, το παιδιατρικό πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται και από ε, άλλες δράσεις και να το βλέπουμε σε σχέση με την απόφαση του Ιουνίου και το πιλωτικό πρόγραμμα ε, για την πρόσβαση στα φάρμακα. Έτσι είναι ευρύτερο πλαίσιο. Διότι ο παιδιατρικός κανονισμός είναι ένα εργαλείο σημαντικό μεν αλλά συγκεκριμένο. Επίσης προσπαθούμε να αναπτύξουμε διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό. Τέλη Σεπτεμβρίου ε, ξεκίνησε μια συνεδρίαση ε, με εκπροσώπους τη FDA των ΗΠΑ, του δικού μας ΕΟΦ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει μια διατλαντική συνεργασία και να υπάρχει και επιπλέον έτσι, χώρος. Γιατί όπως είπατε ε, το πρόβλημα είναι ότι είναι μικρή, μικρό το δείγμα του πληθυσμού με σπάνιες οι ασθένειες ε, κτλ. Ε, πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνατε τώρα και εσείς για την ογκολογία, τους παιδικούς, παιδιατρικούς καρκίνους. Ε, το αναλύσαμε και αυτό με τους αρμόδιους συναδέλφους και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά μπορούμε να δώσουμε άδεια για 11 φάρμακα τα τελευταία χρόνια στην ογκολογία, αντικαρκυνικά. Καλά, δεν είναι και κανένα τεράστιο αριθμό, αλλά πριν ε, το κανονισμό αυτό κυκλοφορούσαν τρία αριθμό, τρία φάρμακα. Ε, βέβαια, η εικόνα είναι πολύ πιο περίπλοκη, ελίμονο. Και θα το λάβουμε υπόψη και στην τελική μας έκθεση. Και μόλις ε, καταρτιστεί θα σας την υποβάλουμε και σε εσά και στο Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θυμίζω μόνο την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 10 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία εδώ στην ΕΜΒΗ θα γίνει στις 8 συγγνώμη, Δεκεμβρίου. Εξαντλήσαμε την ημερησία διαταξή μας. Επόμενη συνεδρίαση 21 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Έκτακτη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λήξη συνεδρίαση.